Ναι, ξεκινάμε αμέσως τις εργασίες μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις αποφάσεις ακριβώς που υιοθέτησαν οι συντονιστές χθες. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι συντονιστές για την ετήσια έκθεση των Ombudsman για το 2010, την Ευρωπαϊκή αυτή χρονιά, να μην ε, αναθέσουν σε κανέναν βουλευτή την έκθεση αυτή, αλλά στην Προεδρία. Και μετά η επόμενη πήγε στους πράσινους και η γνωμοδότηση για τη στρατηγική της ε, Ευρώπης για την ευμάρεια των ζώων 2012-2015 ε, την πήρε το CNSD και επίσης οι συντονιστές προχώρησαν σε μια ανταλλαγή απόψεων για τις αντιπροσωπείες και τις επισκέψεις το 2010 και ακούσαμε τις διάφορες υποδείξεις για Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και τις προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων για να ξεκινήσουμε αυτές τις δραστηριότητες μας και να οργανωθούμε και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν οι συντονιστές θα αποστείλουν στην Προεδρία τις προτάσεις τους για τις επισκέψεις και μετά η Γραμματεία θα αναλάβει τη σύνταξη ενός καταλόγου. Και οι συντονιστές το Μάρτιο στη συνάντησή τους θα αποφασίσουν για αυτό το έγγραφο. Ορισμένες δυνατότητες έχουμε, Ισπανία, Γαλλικία, ας πούμε, και Ελλάδα, Ιταλία κλπ. Και όσον αφορά για τη γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας για τις νέες αναφορές, εκεί δεν πήραμε ακόμα κάτι στα χέρια μας, καμία ανακοίνωση σχετική. Και όσον αφορά τις αναφορές για το Σμόλενγκ, για την αεροπορική καταστροφή, η απόφαση αναβλήθηκε. Θα συζητήσουμε για την πολυναλλευτική πολιτική σήμερα, ξεκινώντας από το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Αυτό έχει να κάνει... Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ε, κάτι που ε, έχει να κάνει λίγο με το θέμα των ε, συντονιστών είναι ότι η Γραμματεία μας έχει στείλει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης ε, για το Μάρτιο όπου υπάρχει η ετήσια έκθεση του 2011 της Επιτροπής μας. Αυτό συνήθως δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως έχω ενημερωθεί σωστά, τότε ασχολούμαστε ακόμα με την ε, καταγραφή και συζήτηση αναφορών από το 2011. Ε, εργαζόμαστε ακόμα με βάση ε, τις αναφορές του 2011. Παρακαλώ λοιπόν να διαγραφεί από την ε, ημερήσια διάταξη του Μαρτίου η ετήσια έκθεση και να τεθεί στην ημερήσια διάταξη όταν έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Αλλιώς μπορεί να έχω ενημερωθεί λάθος, αλλά παρακαλώ να αναβληθεί από το Μάρτιο η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Έχουμε την ε, προέλευση το... και τα θέματα των ε, αναφορών του 2011. Υπάρχει ακόμα λίγη καθυστέρηση όσον αφορά το ποιες έγιναν ε, παραδεκτές. Αλλά ο κύριος Τσίτσεστερ έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεσης με τα βασικά θέματα και νομίζω ότι Θέλει πολύ να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω στην έκθεση αυτή τον Μάρτιο. Βέβαια, οι στατιστικές θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ε, ανάλυσης των θεμάτων αυτών από τα μέλη της Επιτροπής. Ε, Εντάξει, περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Σήμερα το πρωί θα εξετάσουμε τις αναφορές για την αλλιευτική πολιτική. Έχουμε την 10 με δύο αναφορές. Την 860, μάλλον την 802 του 2011 της κυρίας Ανούκ Ντελαφορτρή για την κοινή αλληλευτική πολιτική, η κυρία είναι εδώ παρούσα, και την 860 του 2011 του Πολ Κίντ σχετικά με τις ποσοστώσεις αλίευσης και την υπεραλίευση και έχουν προσκληθεί και μέλη της Επιτροπής Αλίας, όπως επίσης και από Εθνικά Κοινοβούλια. Και το λόγο έχει η κυρία Νούκ Ντελαφορτρή. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσετε εδώ σήμερα για να παρουσιάσω την αναφορά του ΒΒΕΦ. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ σύντομο βίντεο που θα εξηγήσει το πρόβλημα.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 Um, μια πολύ σύντομη εισαγωγή για να σας δείξω περί τίνος πρόκειται. Εμεί ξεκινήσαμε, ανάλαβαμε μια τέτοια πρωτοβουλία για περισσότερα ψάρια πριν από μερικού μήνε σε πολλά κρατημέλη, από πολλά από τα γραφεία μα. Το πρόβλημα τη υπεραλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η υπεραλήψη ουσιαστικά είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τους ωκεανούς μας. Σήμερα 75% των ε, ηχθειακών αποθεμάτων ε, τη χάνουν υπερεκμετάλλευσης, 3 στα 4 δηλαδή, και έως και 60% όλων των αλλιευμάτων πετώνται ξανά στην ε, θάλασσα, είτε νεκρά είτε σχεδόν νεκρά, γιατί συχνά οι αλληλείς δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά είναι και υπερβολικά τεράστιο κόστος ε, προς την κοινωνία. Ε, συνεχώς εξαρτώμεθα περισσότερο από τις εισαγωγέ, καθώς αυτή τη στιγμή 60% όλων των ε, θαλασσινών εισάγονται. 30% των ε, θέσεων εργασίας στον τομέα της αλίας χάνονται κάθε χρόνο και έχει και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος όλο αυτό. Ε, εκτιμούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει 3 δις ευρώ κάθε χρόνο ε, από διαφυγόντα κέρδη ουσιαστικά, ε, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την αλία. Υπάρχουν και λύσεις βεβαίως. Εμείς ζητούμε από τον κόσμο να υπογράψει μια αναφορά σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσει την από πάνω προς τα κάτω βραχυπρόθεσμη διαχείριση ε, και ότι ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα διαχειρίζονται ε, και θα διασφαλίζουν την ε, επιβίωση των, της αλληλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να σταματήσουμε και τη σπατάλη των αλλιευμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, ούτως ώστε οι αλληλείς να αλλιεύουν μόνο ό,τι είναι απαραίτητο και όταν είναι απαραίτητο. Και τέλος, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πολύ σημαντική αλευτική δύναμη ανά τον κόσμο και έτσι όλοι οι κανόνες που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά σκάφη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ισχύουν και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι λύσεις είναι εφικτές αν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Βεβαίως κάποιος μπορεί να διαρωτηθεί ποιος ενδιαφέρεται για την υπεραλίευση. Πέρυσι το ΒΒΕΦ έκανε μια ανεξάρτητη δημοσκόπηση σε 14 κράτη-μέλη και μας εξέπλησε θετικά το, το αποτέλεσμα. 88% των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν τα αλλιεύματα που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προέρχονται από βιώσιμα αποθέματα, δηλαδή που δεν τη χάνουν βεραλίευσης. Και 78% των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, για να διασφαλίσουν ε, μια θετικότερη εξέλιξη. Γι' αυτό και μετά από αυτή τη δημοσκόπηση αποφασίσαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να εκφραστούν, να εκφέρουν την άποψή τους. Πάνω από 57.000 άτομα την έχουν υπογράψει. Αυτό έχει γίνει με εκδηλώσεις στο δρόμο, στην, ε, και στη Σκωτία και στις Βρυξέλλες, βλέπετε εδώ πέρα φωτογραφίες, ε, και μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποια από, τα γραφεία μας ε, τώρα αρχίζει όλη η διαδικασία, αλλά ήδη έχουμε από την Ελλάδα, το Μένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία κτλ. Και ελπίζουμε ε, να λάβουμε αναφέροντος, να έχουμε αναφέροντος από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον 500.000 υπογραφές μέχρι το Σεπτέμβριο, όταν το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα ψηφίσει την αναφορά στην Ολομέλεια βέβαια σε καλύτερη θέση για να εξηγήσει γιατί υπέγραψε αυτή την ε, αναφορά είναι ο Ραούλ που ήρθε από την Ισπανία και ήθελε να εξηγήσει προσωπικά στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί υπέγραψε την αναφορά. Ραούλ, θα μιλήσει ισπανικά. Καλημέρα σε όλους. Ραούλ, από τη Σεβίλη είμαι και θα σας πω μερικά πράγματα. Το μήνυμα σαν ένας πολίτης που υπέγραψε αυτή την αναφορά. Από όταν ήμουν μικρός θυμάμαι ότι πολλές νύχτες του καλοκαιριού ε, ήθελα να υποφεληθώ από την παλήρια και από την αλίευση και πώς άνθιζε η ζωή μετά, φαινόταν η ζωή ε, στην άμποτη. Εδώ λοιπόν πολλές φορές ε, με συγκίνησε και ε, ήθελα να σπουδάσω βιολογία και ειδικευμένο στη θάλασσα και θα ήθελα να σας πω ότι πολλές ε, γεύσεις εξαφανίστηκαν ενώ εξαντλήθηκαν οι αλευτικοί πόροι γιατί πολλές φορές ξεχάσαμε την παραδοσιακή αλίευση, την αφήναμε στην τύχη της και μια βασική δραστηριότητα των ανθρώπων που ζουν σε παράκτιες περιοχές. Ε, τέλειωσε η δραστηριότητά τους, έληξε γιατί δεν υπήρξε κατάλληλη πολιτική για να ταινίσουν το μέλος. Εάν έχω μια οικογένεια θα μπορούσα να πω στους απογόνους μου ότι μία μέρα οι λαοί της ε, ακτής ε, αλίευαν κάποτε και υπήρχαν και πολλές γιορτές, πολλές εκδηλώσεις ε, με αφετηρία τη θάλασσα. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με την εξάντληση των αλλιευτικών πόρων ε, όταν ε, έχω μια δουλειά. Με λυπεί να βλέπω ότι σιγά σιγά υπάρχει μια φθήνουσα πορεία και αναγκάζομαι την εγκαταλείψω. Και εάν δεν ληφθούν μέτρα η Αντζούγια και άλλα πολλά μικρά είδη επίσης βλέπουμε ότι εξαλλαλούνται γιατί δεν προστατεύονται. Εδώ ναι, από δικής μας πλευράς ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε και αν καταβάλουν προσπάθειες θα απαντήσει, θα ανταποκριθεί κατάλληλα και η θάλασσα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και αυτές τις μέρες εμείς ε, υποστηρίχτηκαμε από χιλιάδες ε, πολίτες για να μπορέσουμε εδώ να σχεδιάσω μια νέα αλλιευτική πολιτική του 21ου αιώνα δίκαιη που να σέβεται τη θάλασσα και τους αλείς και που είναι υπεύθυνοι για να σεβαστούν αυτές τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να πούμε τι σημαίνει η θάλασσα για μας, οι συνήθειες, η τέχνη της αλληλείας, οι μορφές ζωής, το είδος ζωής των πληθυσμών αυτών Παντού υπάρχει αλευτικός στόλος ευρωπαϊκός. Είμαστε μεγάλη δύναμη αλληλευτική και περισσότεροι ζητάμε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση και να ε, μας τροφοδοτούν με είδη που να συνεχίσουν να διατηρούνται και εσείς θα μπορούσατε να επηρεάσετε την κατάσταση και στις ευρωπαϊκές θάλασσες αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να μας ξεφύγει αυτή η ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και θα δώσουμε το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο τον κύριο Νίλσεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή πέρυσι πρότεινε να πακέτο σχετικά με την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής για ένα νέο βασικό κανονισμό, για μια νέα ε, οργάνωση της αγοράς, της ενιαίας αγοράς και ανακοίνωση ε, για την ε, διάσταση και το Δεκέμβριο επίσης μια πρόταση για ένα νέο ε, ταμείο αλίας η Επιτροπή βλέπει την αναφορά της ε, ΒΒΕΦ ως ε, μια κίνηση στήριξης ε, της πρωτοβουλίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ από την Επιτροπή. Η αναφορά επιθυμεί όλες αυτές τις αλλαγές που προτείνει και η Επιτροπή στο πρόγραμμά τη. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η υπάρχουσα ΕΚΑΒ δεν ε, έχει λειτουργήσει αρκετά καλά για να επιλύσει τα προβλήματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όπω ε, η υπεραλίευση, η υπερβολική ικανότητα στου στόλου, ε, οι ισχυρέ επιδοτήσει και η μείωση του όγκου των αλλιευμάτων που προκαλείται από του Ευρωπαίου αλλοίς. Γι' αυτό και η Επιτροπή πρότεινε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ελπίζουμε να επιφέρουμε τις αλλαγές που απαιτούνται για την ανατροπή της ε, υφιστάμενης κατάστασης και τάσης ε, στην Αλία. Και η μεταρρύθμιση αυτή θέλει να διασφαλίσει ότι οι Αλίες ε, θα έχουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες συνθήκες για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην διαθεσιμότητα των τροφίμων. ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της ε, αναφοράς που μπορούμε να βρούμε και στην πρόταση μεταρρύθμιση. Έχουμε το ζήτημα της μακροπρόθεσμης διαχείρισης. Ήδη τώρα υπάρχουν αρκετά πολιετή σχέδια για διαφορετικά ηχθιακά ε, ε, από και το θέμα είναι να έχουμε ακόμα μεγαλύτερα τέτοια ε, προγράμματα που να περιλαμβάνουν περισσότερα από θέματα και θα βασίζονται στο στόχο ε, της μεγαλύτερης βιωσιμότητα των αποθεμάτων μέχρι το 2015. Πολύ φιλόδοξο αυτός ο στόχος. Άλλο τμήμα της μεταρρύθμισης είναι ε, η απαγόρευση της, της απόρριψης των αλλιευμάτων στη θάλασσα. Αυτό πάντα προοδευτικά θέλουμε να γίνει, ξεκινώντας από το 2014. Και υποχρέωση θα ισχύει για διαφορετικά αποθέματα. Παρομοίω και για την υπερβολική ικανότητα των στόλων υπάρχει μια νέα προσέγγιση, δηλαδή θέλουμε να προτείνουμε τις, τη δυνατότητα μεταφοράς ε, δικαιωμάτων, ε, αλληλευτικών δικαιωμάτων, γιατί έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ε, για την χρηματοδότηση των σχεδίων παροπλισμού σκαφών και από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργούν σωστά. Και τώρα αυτό είναι ένα νέο μέσο για να καταπολεμήσουμε τον υπερβολικό αριθμό σκαφών ουσιαστικά. Μετά, Άλλο σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η πτυχή της ε, περιφερειοποίησης. Ήδη από τώρα, σε πολλά από τα πολιετή ε, προγράμματα υπάρχει μια τέτοια περιφερειακή προσέγγιση, ε, εστιάζοντας την προσοχή μας σε διαφορετικά αποθέματα, σε διαφορετικές περιοχές. Θέλουμε να τονίσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την πτυχή και στο πλαίσιο και της συνθήκης ε, να μεταφέρουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς τα ενδιαφέρομενα μέρη με συμμετοχή και των αλλιέων σε περιφερειακό επίπεδο για να γίνεται χρήση και να αξιοποιείται και δική τους γνώση κατά τη λήψη και εφαρμογή μέτρων ε, για την ελεία. και θα πρέπει να συμμετέχουν και μεγαλύτεροι ε, αλληλευτικοί φορείς. Μια άλλη πτυχή που συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά είναι η εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ. Αυτή είναι και η πρόθεση της Επιτροπής. Δηλαδή, οι πολιτικές που ισχύουν στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για αυστηρότερα μέτρα και στόχους ε, διατήρησης να ε, εφαρμόζονται οπουδήποτε υπάρχει αλληλευτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών σκαφών. Τέλος, στο πλαίσιο της ε, πρότασης ε, οργάνωσης της κοινής αγοράς θέλουμε να δημιουργήσουμε και να δώσουμε στους οργανισμούς, στους εθνικούς οργανισμούς ε, τα κατάλληλα εργαλεία για να σχεδιάσουν ε, την παραγωγή τους και να ε, προσαρμόσουν καλύτερα την προσφορά και τη ζήτηση. Η προτάσει τη Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, σε συνάρτηση και με υφιστάμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ελληνία, λογικά και κανονικά θα επιφέρει αυτή τη μεταρρύθμιση που απαιτείται για τη βελτίωση της κατάσταση των ε, ηχθειακών αποθεμάτων. Ευχαριστώ. Ναι, ακούσαμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακαλώ τους συναδέλφους τώρα οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Α, κυρία Άουκεν. yes. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την απάντηση και για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες πολύ βασικές ερωτήσεις. Καταρχήν προς την Κομισιόν. Είναι νόμιμο αυτό που κάνουμε. Μπορούμε να διαπραγματευόμαστε όσον αφορά τη φύση. Τη στιγμή που έχουμε ε, επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις, ε, μπορεί η Κομισιόν και το Συμβούλιο να θεωρούν τα ψάρια εταίρο είναι νόμιμο αυτό που κάνουμε. Να λέμε ότι η επιστημονική ε, εκτίμηση δεν είναι έγκυρη. Και δεν μιλώ για την πρότασή σας, μιλώ για την παρούσα πρακτική. Και η ερώτησή μου προς τους αναφέροντες. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Συμφωνείτε με την πρόταση μεταρρύθμισης. Είναι πολύ σημαντικό ε, το να πετύχουμε βελτίωση εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ντέιβις τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που άκουσα τους αναφέροντες. Νομίζω ότι είναι ωραίο να, ακούμε, να ακούω ως πολύ περιστασιακός ε, επισκέπτης στην Επιτροπή σας ε, να ακούω τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι και η Επιτροπή Αλίας ε, χαίρεται με το θέμα αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι σκεφτόμασταν βραχυπρόθεσμα και ότι οι ε, υπουργικές συναντήσεις κάθε χρόνο ήταν πιο πολύ σαν μονομάχη που υπερασπίζονταν ο καθένας ε, τα δικά του συμφέροντα. Ε, και ο διάβολος φυσικά υπάρχει στη λεπτομέρεια. Ξέρουμε ότι η ε, Επιτροπή έχει παρουσιάσει την πρότασή της. Θέλει πολιετή ε, προγράμματα διαχείρισης ε, για όλα τα αποθέματα, ακόμα και για τα δύσκολα, όπως είναι τα αμυκτά αποθέματα της Μεσογείου. Έχουμε όμως πολύ πενιχρά επιστημονικά στοιχεία στα οποία να μπορούμε να βασίσουμε τα προγράμματα αυτά, κυρίως επειδή τα κράτη-μέλη δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να παρέχουν επιστημονικά στοιχεία. Είναι λοιπόν αμφισβητήσιμα τα όρια που θέτει η Κομισιόν για να πετύχει βιώσιμη αλληλεία και να μπορούμε να έχουμε το, την, την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Κομισιόν ε, τι ακριβώς εννοεί. Εννοεί πράγματι τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ή ε, εννοεί την αποκατάσταση της βιομάζας, κάτι που δεν μπορούμε να πετύχουμε μέχρι το 2015. Ε, προφανώς αυτή η συζήτηση είναι που διεξάγεται στην Επιτροπή Αλληλείας. Θα θέλαμε όμως περισσότερα στοιχεία από την Κομισιόν. Και τίθεται το ερώτημα πώς μπορούμε να μειώσουμε την ε, υπερβολική αλλιευτική ικανότητα. Πώς μπορούμε να ε, εμποδίσουμε τα υπερβολικά πολλά πλοία να αλλιεύουν ε, τα λίγα ψάρια που έχουν απομείνει. Έχουν αναφερθεί κάποια προγράμματα παροπλισμού πλοίων τα οποία ε, δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους ε, και γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει μεταβιβάσιμες ε, αλλιευτικές παραχωρήσεις, πράγμα, θέμα επίμαχο. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα μέσο το οποίο θα, θα, θα είναι γενικό, θα καλύψει τα πάντα. Αλλά ένα πρόγραμμα τα μεταβιβάσιμων αλλιευτικών παραχωρήσεων μπορεί να διαμορφωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ε, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα. οι αλληλείς θέλουν ε, δικά τους τοπικά προγράμματα, κάτι που σημαίνει ότι τελικά θα μπορούν να κατηγορούν τους δικούς τους τοπικούς πολιτικούς αντί για τις Βρυξέλλες για την αποτυχία. Τέθηκε το θέμα των απορρίψεων. Ε, ε, το 60% μου λέτε των ηχθείων απορρίπτονται, από αλληλείς έχω ακούσει το 80% λόγω της έλλειψης επιλεκτικών αλλιευτικών εργαλείων. Οι περισσότεροι που τρώνε ψάρια, που δεν γνωρίζουν τίποτα για την αλληλεία, ε, θα θεωρούσαν ότι όλα αυτά είναι τελείως ε, λάθο, ε, είναι ανήθικα και αποτελεί σημαντική σπατάλη πόρου που μας οδηγεί στην εισαγωγή περισσότερων ψηριών ο καθένας ε, λέει ότι ε, να καταργήσουμε τις, ε, να δώσουμε τέλος ε, στις απορρίψεις, αλλά μόλις μπουν στις λεπτομέρειες λένε ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Αυτή θα πρέπει να είναι η βασική αρχή μας. Αν σταματήσουμε τις απορρίψεις, η πείρα της Νορβηγίας και άλλων χωρών μας δείχνει ότι αν πούμε στους αλείς ότι δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται ψάρια, αυτό δημιουργεί μια δυναμική. Οι άλλοι λένε δεν έχουμε τα επιλεκτικά εργαλεία. Μόλις όμως εφαρμοστεί μια απαγόρευση ε, απορρίψεων, ξαφνικά επινοούνται ή βρίσκονται ε, ή ε, προσαρμόζονται τα επιλεκτικά αλλιευτικά εργαλεία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε τέλος στις απορρίψεις και ε, να μην υπερασπιστούμε από νομικής πλευράς τουλάχιστον ε, τις απορρίψεις. Ε, τώρα αν κάποιος απορρίπτει μεσάνυχτα μέσα στη μέση του ωκεανού αυτό είναι άλλο θέμα. Επικροτώ την αναφορά και ελπίζω ότι και η Επιτροπή Αλληλείας θα επικροτήσει την αναφορά αυτή. Όλοι θέλουμε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά όπως σας είπα, ο διάβολος βρίσκεται σε λεπτομέρεια και τα πολιτικά επιχειρήματα θα περιστρέφονται γύρω από αυτά τα θέματα, τα οποία είναι ζωτική σημασία για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που να μας οδηγήσει σε μια βιώσιμη ελευτική πολιτική για το μέλλον. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Ναι. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Αναφορών που μας κάλεσε να παραστούμε σήμερα εδώ. Δεν ε, θα ξεκινήσω μία συζήτηση. Ακούσαμε πολλά ήδη, αλλά για τους αναφέροντος θα ήθελα να τους καθησυχάσω σας απασχολεί το μέλλον της αλίας και, σε, και εμάς μας απασχολεί το ίδιο. Σας ε, το να διατηρηθούν οι ελευτικοί πόροι και εμάς μας απασχολεί αυτό το θέμα και μας απασχολούν, ε, μας ενδιαφέρουν οι αλίες. Θα πρέπει να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα και εργαζόμαστε στην Επιτροπή Αλίας του Επικοινοβουλίου σκληρά πάνω σε μια μεταρρύθμιση, σε ένα σχέδιο που θα πρέπει να το επεξεργαστούμε ώστε να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα αυτού και Εργάζονται αρκετά πολιτικά κόμματα με διάφορα μέρη. Ο καθένας έχει ένα εισηγητή και εδώ και αρκετούς μήνες προχωράμε, προχωράμε, επαναλαμβάνω, εργαζόμαστε για να πετύχουμε επιτέλους μια νέα και καλή και σωστή μεταρρύθμιση Τη κοινή αλλιευτική πολιτική, Βέβαια πολλά πρέπει να γίνουν και εσείς ε, μπορείτε να βοηθήσετε ιδιαίτερα. Αυτό σας λέω ότι υπολογίζουμε και στη δική σας τη βοήθεια γιατί μαζί σας με όλους θα πετύχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Την επιθυμούμε όλοι μας ε, και για το Ραούλ ε, ναι, και εγώ έχω παιδιά και εγώ θέλω τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μου να βλέπουν μια θάλασσα ανοιχτή μπροστά τους με τους πόρους που επιθυμούμε. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για την ε, συμμετοχή σας. Γιάρν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι εμπειρογνώμων σε θέματα αλληλείας. Ωστόσο, μία συμπληρωματική ερώτηση από την δική μου πλευρά. Ε, έχουμε μια πολύ καλή πολιτική θέση, πολιτική κατάσταση ε, για ε, πολιτική συζήτηση, διότι ακούσαμε την αναφορά και η Κομισιόν λέει ότι α, την αναφορά σας την θεωρούμε ενθάρρυνση να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Προτείνω λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ε, διαδικασία αυτή ε, που ξεκινάει τώρα. Η Κομισιόν ε, δουλεύει, το Κοινοβούλιο λαμβάνει αποφάσεις. Η δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση από πλευράς μου είναι... Ο τίτλος πράγματι είναι σωστός. Όλοι θέλουμε τα ίδια, όλοι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Ποιο είναι ο τομέα ε, στην αναφορά σας που πιστεύετε ότι υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για ε, βελτίωση και πού πιστεύετε ότι ε, οι απαιτήσει και η πραγματικότητα απέχουν περισσότερο η μία από την άλλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Μέρ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τους αναφέροντες και μπορούμε τώρα να συζητάμε μαζί τους για την πολιτική, την αλληλευτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άποψη της ομάδας μου συμφωνεί σχεδόν με όσα υπόθηκαν από τους αναφέροντες. Για μας είναι σημαντικό να υπάρξει μια εγγύηση ακριβώς και να βοηθήσουμε για τους αλευτικούς πόρους και θα πρέπει να έχουμε μια υφόρο ανάπτυξη για να συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα με θέσεις απασχόλησης ποιοτικές και με εγγύησεις επίσης για προμήθεια ε, θα ήθελα να πω κάτι το γενικό για την αλία, την ερασιτεχνική και γιατί έχει, να κάνει, έχει μεγάλη σχέση με την ε, για εκατοντάδες χρόνια ε, συνήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αλία που να μπορεί να συνεχιστεί και να σέβεται και τη φύση. Για μας λοιπόν οι σκέψεις αυτή είναι θετική για να ε, επιδιώξουμε την αηφορία και μια κοινή αλληλευτική πολιτική που θα εγγυηθεί τις θέσεις απασχόλησης και η έρευνα να τεθεί στην υπηρεσία αυτής της αηφορίας, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και κρατικά και κοινοτικά και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την αναφορά. Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει επίσης, λέω και εγώ, να παραμείνει ανοιχτό το θέμα στην αναφορά αυτή. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία... Συγγνώμη, επειδή το ξέχασα πριν ε, στις ε, ερωτήσεις μου, τον αντίκτυπο της ρήπανσης ε, και από τις ρήπανσεις από το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στις εκτιμήσεις. Γιατί Έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα για την ε, επίπτωση του Διευθυντήτου του άνθρακα στα κτηριακά θέματα. Ναι. Από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής θα ήθελα να ζητήσω μήπως θέλει να απαντήσει κάτι να Ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο ερώτημα που θέσατε, Δηλαδή αν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τη φύση. Και αν η Επιτροπή παρακάμπτει τις ε, επιστημονικές νοματεύσεις ήδη τώρα, οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται στα ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό είναι προφανές στις προτάσεις της Επιτροπής. Το ζήτημα είναι ότι δεν μιλάμε για θετική επιστήμη εδώ πέρα, δεν μπορούμε ακριβώς να μετρήσουμε τον αριθμό των ψαριών. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία κινδύνου ε, κατά την ε, κατάρτιση τέτοιων σχεδίων για την αλία. Μπορούμε όμως να βασίσουμε τις ε, πολιτικές μας στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές νοματεύσεις και να ελπίσουμε ότι ακολουθούμε αυτές τις συμβουλές στην εφαρμογή των πολιτικών. Ο κύριος Ντέιβις ε, έκανε ορισμένες παρατηρήσεις ε, για την ε, πρόταση μεταρρύθμισης. Περισσότερο παρατηρήσεις παρά ερωτήσεις. Πράγματι, Υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων για αρκετά από αποθέματα και εκεί η Επιτροπή προτείνει η συλλογή δεδομένων να, ότι πρέπει να, να, βελτιωθεί, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί ε, αυτή η δραστηριότητα και ότι εκεί που δεν υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα, αυτό να μην αποτελεί ε, δικαιολογία για να μην ε, λαμβάνονται τα μέτρα για να καταστεί βιώσιμη η αλεία. Αυτό είναι το τμήμα της πρότασης. Μετά για το MSY και το BMSY. Ε, μπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα, όμως νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση. Πράγματι, μέχρι το 2015 θα είναι δύσκολο να αποκαταστήσουμε το BMSY. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να πάμε στο FMSY και μετά μακροπρόθεσμα στο BMSY. Ε, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να είμαστε λίγο πάνω από το MSY, γιατί ε, τα αποθέματα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ε, και υπάρχει μια, ένα περιθώριο, αν θέλετε, και αν έχουμε έναν στόχο που είναι λίγο πάνω από το MSY, θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Θα έχουμε και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να είμαστε πιο κοντά στο MSY και να μην ε, υπάρχουν διακυμάνσει πολύ κάτω από τον στόχο. Τώρα για την ε, υπερβολική ικανότητα, αλληλευτική ικανότητα, είναι σημαντικό να, να υπογραμμίσουμε αυτό που είπε ο κ. Ντέιβις, ότι ε, πολλά λέγονται για αυτό το, μέσο της ε, υπερβολικής ικανότητας και ότι μπορούν να, να οικοδομηθούν τέτοια ε, προγράμματα που θα επιλύσουν τις ανησυχίες και θα διασκεδάσουν τις ανησυχίες για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ε, σχεδίων ε, αναχώρα. Γιατί πολλές χώρες, κάθε χώρα χειρίζεται διαφορετικά την κατανομή των ποσοστώσεών της. Όμως πράγματι μπορεί να υπάρχει ένα σωστό σύστημα και έχουμε δώσει αυτή την ελευθερία στα κρατημέλη να φτιάξουν δηλαδή το σύστημά τους όπως επιθυμούν. Και αυτό παρέχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να διασκεδάσει τις ανησυχίες ε, ορισμένων κρατομελών. Επίσης, για, την, για τις απορρίψεις και πάλι είναι δύσκολο να το ε, εφαρμόσουμε, ιδιαίτερα ε, στα, στην ανάμεικτη αλληλεία, αν θέλετε, γιατί πολλές φορές έχουμε ανάμεικτα αποθέματα που αλλιεύονται. Όμως και πάλι σημαντικό να θέσουμε ένα στόχο της μείωσης και κατάργηση των απορρίψεων, γιατί αυτό ε, συνδέεται και με την, ε, με την επιλογή αποθεμάτων. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που θέσατε. Υπήρχε και το τελευταίο ζήτημα του αντικτύπου της ρήπανση στα αποθέματα. Εγώ δεν είμαι ειδική στην ΕΛΗ, e, αλλά είναι προφανές ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν ε, την κατάσταση των θαλασσών και ένας από τους ε, παράγοντες ε, που ε, συμβάλλουν στην κατάσταση, στη σημερινή κατάσταση είναι και η αλία, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εξίσου σημαντικοί. Είτε μιλάμε για, για τη ρήπανση, είτε το άνθρακα, την αλλαγή της θερμοκρασίας στη θάλασσα που οδηγεί και στην αλλαγή των μεταναστευτικών ροών των νυχθείων. Όλα αυτά τα πειράζουν, αλλά βεβαίως και η αλία είναι σημαντικός παράγοντας. Σας ευχαριστούμε. Και για να ολοκληρώσουμε, εάν κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο από τους συναδέλφους, ε, θα ήθελα να ζητήσω από την υπογράφουσα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω μία σύντομη απάντηση και για την ε, πιο μακροσκελή απάντηση να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ρομπέρτο Φερίνιο. Η σύντομη απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Άουκεν είναι τι γνώμη έχουμε για την πρόταση της μεταρρύθμισης. Πιστεύουμε ότι είναι καλή, έχει καλά στοιχεία, αλλά όπως ανέφερε ο κύριος Ντέιβις, ο διάβολος ε, υπάρχει στη λεπτομέρεια και ελπίζαμε ότι η ίδια η πρόταση θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη με την έννοια ότι πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό με την ποικιλία αλληλείας που υπάρχει στην Ευρώπη. Ε, συχνά δεν υπάρχει ε, μία γενική λύση που μπορεί να ισχύει για όλους, όπως για παράδειγμα στο θέμα των απορρίψεων. Θα θέλαμε λοιπόν η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αλλιέων, ε, θα μπορούσε να δώσει την καλύτερη απάντηση για, τις, για τους διάφορους τύπους στην Ευρώπη και ελπίζαμε ότι θα δούμε περισσότερα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων για την συνδιαχείριση της αλληλείας στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να ε, ψηφίσει πάνω στο θέμα της, ε, της αλληλείας και της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Είχαμε τρεις αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν που στόχο είχαν ε, την βιώσιμη αλληλεία και την εξάλληψη της υπεραλίας. Ε, είναι μια μοναδική ε, ε, περίπτωση διότι το 2022, την επόμενη φορά δηλαδή, κανένα απόθεμα δεν θα βρίσκεται σε βιώσιμο επίπεδο. κινδυνεύουμε λοιπόν να χάσουμε όλα μας τα αποθέματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα πρέπει να αποσχολεί την Επιτροπή Ελίας αλλά και όλους τους βουλευτές, το να σώσουμε τους ωκεανούς και επίσης θα πρέπει να έχουμε ηγετική θέση παγκοσμίω, διότι η ευρωπαϊκή αλληλεία σημαίνει πολλά και για την Αφρική και για την ε, Ασία. Διότι εκεί μας λένε ε, ότι δεν είναι ότι μας εκμεταλλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λένε. Ε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει μια βιώσιμη ημερήσια διάταξη, ένα βιώσιμο θεματολόγιο παγκοσμίω. Ε, τα ασιατικά κράτη θέλουν πρότυπα ε, στα οποία να μπορούν να ε, προσφεύγουν. Κατά τους επόμενους μήνες απομένει πολλή δουλειά για το Κοινοβούλιο να βελτιώσει και να εκπονήσει τις λεπτομέρειες για να δοθεί τέλος στις απορρίψεις και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Ναι, αυτή ήταν η σύντομη απάντηση. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφο ε, Ρομπέρτο Φερένιο θέλει κάτι να προσθέσει σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ρομπέρτο Φερένιο, ε, είμαι διευθύντης ε, της πολιτικής μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτική πολιτική του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση στι Βρυξέλλε. Ποια λοιπόν είναι τα μέρη τη πρόταση τη Επιτροπή που μπορούν να βελτιωθούν. κατά τη γνώμη μα, αυτό που έλειπε μέχρι σήμερα είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε τους, τη διαχείριση των ε, φυσικών πόρων. Ε, τα ψάρια αποτελούν μέρος των ωκεανών ε, και όταν μιλάμε για τη διαχείριση φυσικών πόρων μιλάμε για την οικονομική και οικολογική διάσταση και μέχρι τώρα η οικολογική διάσταση απουσίαζε τελείως από την κοινή πολιτική οποιοδήποτε μιλάει εκ μέρους των αλλιέων ε, θα πρέπει να ε, ακούει και το επιχείρημα ότι χάνουμε θέσεις απασχόλησης στον τομέα διότι δεν είναι βιώσιμη η αλλιευτική μας δραστηριότητα. Ε, από οικολογικής και από οικονομικής πλευράς. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το βασικό πρόβλημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να το λύσουμε. Έχουμε έναν βασικό κανονισμό. Η Κομισιόν προτείνει ένα πακέτο ε, μέσων και όπως είπε ο κύριος Ντέιβις, ο διάβολος υπάρχει στη λεπτομέρεια. Και κατά τη γνώμη μας οι λεπτομέρειες είναι οι οικονομικές λεπτομέρειες. Πώς τα οικονομικά μέσα του ε, ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Φύση συνδέονται με τους στόχους του κανονισμού. Και γι' αυτό το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση επιμένει ο κανονισμός να περιλαμβάνει γενικούς στόχους και υποοικονομικούς και υποοικολογικούς όρους και μέχρι τώρα λείπουν οι στόχοι αυτοί. Θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε μια για πάντα να συνδυάσουμε τους, ε, τις οικονομικές και οικολογικές επιτυχίες ε, των ε, αλληλευτικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα, διότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις ε, διαπραγματεύονταν την κατανομή οικονομικών μέσων πίσω από κλειστέ πόρτες. Πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση αυτού του μηχανισμού. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε την διαχείριση των φυσικών πόρων και θεωρούμε την την ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, ως διαδικασία παράλληλη με την ε, οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική για να πετύχουμε καλή κατάσταση του ωκεανού μας μέχρι το 2020. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα, συνδυασμένα και θα πρέπει και πάλι να συνδυάσουμε το, την οικολογική και οικονομική διάσταση. Ευχαριστώ. Προτείνω λοιπόν να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά αυτή. Να τη συζητήσουμε και πάλι το Μάιο όταν θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την αλλιευτική πολιτική. Σημαντικό είναι να μπορέσουν να συμμετάσχουν πολίτες μαζί με μέλη της Επιτροπής Αλίας. Στη συνάντηση του Μαΐου θα εξετάσουμε παρόμοιες αναφορές στα πλαίσια της εκστρατείας Fish Fight, μάχη για την αλία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε τις εξής αναφορές. Την αναφορά 295 του 2009, Des May, Ιρλανδικής Ιθαγένειας, για τον αποκλεισμό των αλλιέων από τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος διαχείρισης του χελιού για την Ιρλανδία. Επίσης, την 909 του Ζαν Πολ Ντορόν, γαλλικής ηθαγένειας, εξ της Γαλλικής Εθνικής Ομοσπονδίας Αλίας για το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης για τη διατήρηση των αποθεμάτων χελιών. Επίσης, την 754 αναφορά του 2011 του Σαλβαντόρ Πιερό Γκόμεθ ισπανικής Ιθαγένειας ε, για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού και για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Ε, κανείς όμως από τους αναφέροντες δεν είναι παρόν, γι' αυτό παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στα συμπεράσματά της. Ο κ. Θεοφίλου και ο συναδελφός του. Mr. O'Shea. Good morning. Good Καλημέρα. Πάντα ονομάζομαι. Εκπροσωπώ την Επιτροπή. Είμαι, συγγνώμη, από την Δυτική Ένωση Αλλιέων. από τη Western Eel Fishermen Association. Υπάρχουν ε, προϋποθέσεις ε, που καθορίζονται στον ε, κανονισμό 11, 11.00 του 2007. Η φύση του κανονισμού μας δείχνει Ποιε ε, ε, δραστηριότητε θα πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο της επικουρικότητα, ε, λαμβάνοντα υπόψη και τι τοπικές ιδιαιτερότητες. Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι ο οικονομισμό απλώ περιγράφει τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν, δηλαδή την ανάκαμψη των αποθεμάτων, αφήνοντας 40% των χελιών να ξεφύγουν. Και μα οδηγεί στην απόφαση ε, μάλλον το πώ θα γίνει αυτό, το πώς επιτευχθεί ο στόχος, είναι ζήτημα του κράτους μέλους. Το κράτο μέλος επιλέγει τα μέσα για την επίτευξη του στόχου. Η Ιρλανδία έχει επιλέξει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχει αξιολογήσει η ISIS ε, στο πλαίσιο και του ε, Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης για τα χέλια. Και από όσο γνωρίζει η Επιτροπή, η Ιρλανδία έχει διαβουλευθεί τους, με ε, με τα διαφέρμενα μέρη σε δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα το 2008. για να Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί προεδρεύω μιας συνεδρίασης. αλλά έχω κάποια εμπειρία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε και είχαμε πολλές ε, παρουσιάσεις ε, μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούσαν εκείνες τις περιοχές. Βεβαίως και υπάρχει ζήτημα επικουρικότητας και λαμβάνονται τα απαραίτητα ε, μέτρα, όμως καθυστερήσαμε, υπήρξε καθυστέρηση ε, για να δώσουμε το λόγο στα πραγματικά ενδιαφέρομενα μέρη. Γιατί οποιαδήποτε μείωση της ποσοστώσης ε, επηρεάζει πάνω απ' όλα όχι τη βιομηχανία ή το κοινοβούλιο, του πολιτικού, αλλά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και λάβαμε 16 υποβολές ε, ε, ως απάντηση στην πρόσκληση του κοινοβουλίου. Και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μην τους καλέσαμε, μπορεί να μην είχαμε καλέσει καθόλου, Απλώς είχε ξεκινήσει η δικασία εδώ και καιρό και λειτουργούσε σωστά. Ίσως δηλαδή από νομικής πλευράς ε, να εκπληρώθηκαν όλες ε, οι προϋποθέσεις, αλλά υπήρχαν και ηθικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν. Γι' αυτό και συμφωνώ ότι θα πρέπει να το επαναξετάσουμε, γιατί εν τω μεταξύ δεν υπάρχει αλίευση χελιού. Αλλά θυμάμαι πριν από πέντε χρόνια ότι η Ιρλανδία Λύης διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπαν ότι σε 19 χρόνια θα μπορούσαμε να το επαναξετάσουμε αυτό. Τώρα, εντάξει, δεν είμαι πολύ τόσο ενήμερος, αλλά νομίζω ότι έχουμε αργήσει υπερβολικά, γι' αυτό θα πρέπει να το επαναξετάσουμε εκ νέου. και ελπίζουμε να συνάδουμε και με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠΚΙ το 2014. Βλέπω εδώ και τον ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Αλίας και το, το ένα... Το ένα σύστημα που να λειτουργεί για όλους, αυτό δεν λειτουργεί. Πρέπει να υπάρχει περιφερειοποίηση και επικουρικότητα. Γι' αυτό και θα πρέπει να το επαναξετάσουμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστούσουμε. Κανείς άλλος δεν ζητεί το λόγο, γι' αυτό από πλευράς Επιτροπής ε, μήπως μπορείτε να απαντήσετε για τον κύριο Γκάλαχερ. Good morning. Uh, I'm... Καλημέρα σας. Λέγομαι Χρήστος Θεοφίλου. Είμαι συνάδελφος του Μπρένταν και συντονίζω οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χέλια εντός της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Θα προσπαθήσω λοιπόν σύντομα να απαντήσω σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που μόλις έγιναν. Είναι αλήθεια ότι υπολογίζεται ο χρόνος αποκατάστασης σε 19 χρόνια. Μπορεί αυτό να ακούγεται ε, ακραίο. Μπορεί να ακούγεται σαν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση των χελιών, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουν μεγάλο χρόνο αναπαραγωγής τα ε, χέλια. Ανάλογα με τις περιοχές ε, μπορεί να χρειάζονται πάνω από 20 χρόνια να αναπαραχθούν. 19 χρόνια λοιπόν είναι τέσσερις γενιές, που δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα για την αποκατάσταση. Ευτυχώς όμως εντός του κανονισμού έχουμε μία διάταξη στο άρθρο 9 όπου λέει ότι τα κράτη-μέλη απαιτού... Ε, απαιτείται από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν έκθεση πρόοδου μέχρι την 1η Ιουλίου φέτος. Σε λίγους μήνες δηλαδή. Ήδη έχουμε ετοιμάσει έναν πίνακα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη κατά την προετοιμασία των εκθέσεων και η Κομισιόν Μέχρι το 2013 θα έχει εξετάσει όλες τις εκθέσεις αυτές και θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια γενική έκθεση πάνω στην ε, πρόοδο που θα έχει σημειωθεί ε, με το, την εφαρμογή του κανονισμού για τα χέλια. Όταν λοιπόν θα έχει εξεταστεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο η έκθεση αυτή μπορεί να προτείνουμε τροποποίηση στον κανονισμό, ε, δηλαδή τροποποίηση και στα σχέδια διαχείρισης των κρατών μελών ώστε να διασφαλίσουμε την ε, καλή αποκατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, επιτρέψτε μου να θεωρήσω πολύ σωστή την απάντηση αυτή. Ελπίζω όμως η Κομισιόν να επιμείνει ώστε ε, ε, η αρμόδια υπηρεσία της Ιρλανδίας να υποβάλει την έκθεση μέχρι την 1η Ιουλίου. Υπάρχει, είπατε, πίνακα που μας βοηθεί, αλλά μήπω μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό, να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό μέσα στο επόμενο δεκάμινο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρέμβασή σας. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο τη Επιτροπής, τον κύριο Θεοφίλου, λέει η Πρόεδρος. Αφού συζητήσαμε για τη 295 να μας πει μερικά πράγματα για τις υπόλοιπες δύο αναφορές. Θα προσπαθήσω να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις πολύ σύντομα για να καλύψω και τις δύο αναφορές και μετά να δώσω το λόγο σε όποιον θέλει να πει κάτι πιο συγκεκριμένα. με βάση και τα όσα είπε ο συνάδελφος Μπράντον, ε, αφήνει μεγάλο περιθώριο κανονισμό στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ε, ποια μέτρα θέλουν ε, να εφαρμόσουν για να επιτύχουν τον κοινό στόχο που καθορίζεται στον κανονισμό. Αναπόφευκτα, σε κάθε κράτο μέλο υπάρχει διαφορετική κατάσταση, διαφορετική αλληλεία, διαφορετική ρήπανση, διαφορετικά εμπόδια, παράσιτα, παθήσεις που επηρεάζουν το χέλι. Είναι λοιπόν περίπλοκη και ποικιλόμορφη η κατάσταση, γι' αυτό και επιλέγουμε στα κράτη-μέλη να ε, ε, δίνουμε τη δυνατότητα στα κρατημέλη να επιλέγουν τα μέτρα τους. Κάποια κρατημέλη έχουν επιλέξει ε, μια αυστηρότερη διαχείριση, ενώ κάποια άλλα λιγότερο αυστηρή. Ωστόσο, κάθε σχέδιο υπόκειται σε έλεγχο από την Διεθνή Ένωση ε, Εξερεύνησης των Θαλασσών και από την Επιτροπή. Πριν από την έγκριση κάθε σχεδίου είχαμε πολλούς γύρους με κάθε κράτος μέλος ε, και τους ζητήσαμε να μας παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες ή να βελτιώσουν κάθε πτυχή του σχεδίου και ούτε καθεξής. Για να είμαστε πεπισμένοι ότι κάθε ε, σχέδιο θα επιτύχει τον κοινό στόχο. Συνοψίζοντας, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε συγκεκριμένα μέτρα στα κράτη-μέλη, να τα υποχρεώσουμε δηλαδή να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την αλληλεία ή άλλα μέτρα. Εφόσον επιτύχουν το στόχο, εμάς δεν μας απασχολεί τι μέτρα λαμβάνουν. Δεν έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση. Όχι. Όχι. Άρα λοιπόν ολοκληρώνεται η συζήτηση. Προτείνω οι αναφορές αυτές να παραμείνουν ανοιχτές. Φτάσαμε τώρα στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την 99 του 2011 του Μιγγέλ Σαραγκώσα Φερνάντες, Ισπανικής Ιθαγένειας, σε μια, σχετικά με μια παραδοσιακή επιλεκτική αληφτική τεχνική, την Μπονιτολέρα στα Ισπανικά. Απόν ο αναφέρον, άρα λοιπόν εκπρόσωπος της Επιτροπής, η κυρία Μπάρμπαρα Φοκέτ, έχει το λόγο η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, Barbara Φόκε, Desk Officer στη Γενική Διευσιαλία ε, σχετικά με τα θέματα στην ε, Μεσόγειο και κυρίως ε, Γαλλία-Ισπανία. Μέσω αυτής της αναφοράς ο κύριος Φερνάνδες τι ζητάει να αναθεωρήσουμε το παράτημα 2 του κανονισμού για τη Μεσόγειο, γιατί κατά την άποψή του δεν μπορούν να ισχύσουν αρκετές παράκτειες αλλιευτικές δραστηριότητες στην Ισπανία και κυρίως στην περιοχή του Δήμου του. Ο κανονισμός ε, για τη Μεσόγειο ακριβώς έχει να κάνει και με την ε, μικρή παράκτια πολιτική αλλά και παντού στη Μεσόγειο είναι ο πρώτος κανονισμός που ειδικά ειδικά πλαισιώνει κάθε είδους δραστηριότητα αλλιευτική και ε, ο κανονισμός αυτός ε, προβλέπει αρκετή ευλογησία για να μπορέσουν εκεί σε εισαγωγικά να βολευτούν ε, οι διάφορες μορφές αλίας όπως και αληφτικά δίχτυα και άλλα παρόμοια όπως προτείνει και ο αναφέρον. Ζητάει λοιπόν την αναθεώρηση, την διάσταση, της διαστάσεις αυτών των δικτυών στα πλαίσια της Μπονιτολέρα και ε, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά όμως τα μέτρα περιορίζουν έτσι την αλληλεία όπως θα πρέπει και είμαστε ε, υπέρ του να βοηθήσουμε στη Μεσόγειο για να εξασφαλίσουμε μια υφόρο ανάπτυξη και υπεύθυνη αντιμετώπιση αλλιευτική. Θεωρούμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται αυτός ο κανονισμός, το παράδειγμα αυτό να θεωρηθεί, γιατί έστω και αν έχει αγκριθεί το 2006 ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στο σύνολό του μόνο από την 1η Ιουνίου του 2010, γιατί υπήρξαν πολλές και διάφορες ε, Προσωρινέ εξαιρεσει. και πιστεύουμε ότι θα πρέπει πρώτα ειδικά να δούμε πώ ο κανονισμός αυτός συγκεκριμένα εφαρμόστηκε σε κάθε ρυθμισή του πριν να προβλέψουμε μία περαιτέρω μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστούμε. Ναι, σας ευχαριστούμε και εμείς. Μήπως κάποιος τώρα θα ήθελε να λάβει το λόγο σχετικά με αυτό. Όχι. Κανείς. Άρα λοιπόν προτείνουμε να παραμείνει ανοιχτό το θέμα της ε, αναφοράς αυτής. Περνάμε στο σημείο 13 της σημερινής διάταξης. Είναι η 668 του 2011 αναφορά από Γερμανό πολίτη σχετικά με την αλία με ψαροντούφεκο στην Καρσική. Απόν ο αναφέρον ε, προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος. Η κυρία Μπάρμπαρα Φωσέ έχει το λόγο και πάλι. Ναι, και πάλι για να συνοψίσω με λίγα λόγια περί τίνος πρόκειται. Ναι, αναφέρει στην Κορσική παράνομες ενδεχόμενα δραστηριότητες γιατί έχουν να κάνουν με ψαροντούφεκα που είναι άλλο είδος αλίας βάσει του κανονισμού αλίας στη Μεσόγειο. Ο αναφέρον ναι, μας λέει ότι η αλία αυτή πραγματοποιείται, διεξάγεται. Ίσως θα πρέπει να δούμε και πάλι το κείμενο του κανονισμού που λέει ότι αυτή η αλία με ψεροντεύκα απαγορεύεται μόνο αν ε, υπάρχει και, υπάρχουν και μπουκάλες, δηλαδή αν συνδυάζεται με αυτό. Θα πρέπει όμως να απευθυνθεί κανονικά στις γαλλικές αρχές, γιατί ο πρώτος υπεύθυνο για τον έλεγχο της αλίας είναι το κράτος μέλος και η Επιτροπή απλά και μόνο αναλαμβάνει τον εξετάσει εάν τα κράτη-μέλη σέβονται τις ρυθμίσεις της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και ελέγχει αυτές τις διατάξεις και την εφαρμογή και ταυτόχρονα μήπως θα μπορούσε στην Επιτροπή μας να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες που μας χάρη φωτογραφίες που δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται αναπνευστικές συσκευέ, μπουκάλες και ψαροντούφεκα ταυτόχρονα. Και ε, περιμένουμε αυτές τις φωτογραφίες μας λέει ότι με τον ε, τοπικό Οργανισμό Τουρισμού στην Κορσική και με το Βιολογικό Ιστιτούτο ε, ήρθε σε επαφή. Δεν έχουμε ακόμα την απάντηση στα χέρια μας, αλλά εποφελούμε τις ευκαιρίες για να σας ε, αναφέρω τα στοιχεία αυτά και να σας πω ότι στη φωτογραφία, ναι, τελικά μας έστειλε φωτογραφία, αλλά δεν βλέπουμε καθαρά αυτές τις αναπνευστικέ συσκευές μπουκάλες. Ε, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι το συγκεκριμένο, ότι πραγματικά πραγματοποιήθηκε αυτή η παράνομη αλίευση και επίσης θα θέλαμε, επαναλαμβάνουμε από τους αναφέροντες, να απευθυνθούν στο Υπουργείο Αλίας στη Γαλλία που είναι και το αρμόδιο όργανο για την άσκηση αυτού του ελέγχου για την αλία και που θα είναι και ο καταλληλωτός φορέας για να απαντήσει στα ερωτήματα του αναφέροντος. Ευχαριστώ την Επιτροπή για όσα μας διευκρίνησε. Μήπως κάποιος συνάδελφος επιθυμεί το λόγο. Όχι. Και πριν να πάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν της σημερινής διάταξης, προτείνω να παραμείνει ανοιχτό το θέμα αυτό. Πάμε στο σημείο 14 της σημερινής διάταξης. Είναι η 1824 αναφορά του 2009 του Αντώνιο Λόρες Φράνκο εξ ονόμας της πλατφόρμας για την προστασία του κόλπου Σαν Σιμών σχετικά με μια μονάδα παραγωγής ηχθιάλευρου κοντά στο Βίγκο στην Ποντεβέδρα. Απόν ο αναφέρον το λόγο έχει η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής, ο εκπρόσωπος Επιτροπής, ο κ. Ντέβιντ Κρίμον. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Κυρία Σουέμεν, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Αυτή η αναφορά αφορά ένα, ε, μια μονάδα ε, παραγωγής ηχθιελαίου Το κύριο πρόβλημα που αναφέρεται εδώ είναι ότι αυτή η εγκατάσταση δεν θα έπρεπε να έχει λάβει αδειοδότηση το 2008 για τους εξής λόγους δεν υπήρχε η e κα, καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι η υπερβολοντική και η ρήπανση και η ρήπανση του νερού που προκαλείται παραβιάζει το εθνικό δίκαιο βάσει των νόμων που ισχύουν για τα υπόγεια ύδατα σε αυτήν την περιοχή. Τι έκανε λοιπόν η Επιτροπή εδώ. Πρώτον, υπήρξε μια πρώτη ε, γραπτή ανακοίνωση και αποστολή προς ε, την ε, Επιτροπή Αναφοράς το 2010 και έτσι ενημερώσαμε την Επιτροπή ότι υπόγειται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο την EIA και την IPPC σε αυτές τις δύο οδηγίες. Όμως έλαμε περισσότερες ε, πληροφορίες και έτσι ανοίξαμε ένα πιλωτικό φάκελο. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιούμε για να ζητήσουμε επισήμως πληροφορίες και διευκρινήσεις από τα κράτη-μέλη για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. και θίξαμε κάποια ζητήματα στις Ισπανικές Αρχές. Αν υπήρξε τέτοια ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν υπήρξε τέτοια αδειοδότηση IPPC, αν υπήρξαν επιθεωρήσεις. Οι Ισπανικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011 και βάσει αυτών των πληροφοριών η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο τη Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Τουλάχιστον εμεί δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε κάποια παραβίαση. Ε, υπήρξε δεύτερη επιστολή της Επιτροπής προς την Επιτροπή Αναφορών το Σεπτέμβριο, ε, αναγεννώνοντας ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα ε, συγκεκριμένη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Τώρα θέλω να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτο ζήτημα, εάν η οδηγία EIA παραβιάστηκε, η οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να θυμάστε ότι αυτή η εγκατάσταση, αυτή η μονάδα λειτουργεί από το 1976, όταν δεν υπήρχε αυτή η οδηγία. Σήμερα, αυτή η μονάδα πράγματι καλύπτεται από, την, ε, από το δεύτερο παράρτημα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η φυστάμενη μονάδα, τη στιγμή υιοθέτηση της οδηγίας, δεν καλύπτεται από την οδηγία παρά μόνο αν υπάρχουν αλλαγές που επηρεάζουν ή επεκτάσεις που επηρεάζουν την μονάδα και αυτές οι αλλαγές ή επεκτάσεις ε, ε, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Προς το παρόν, οι Ισπανικές αρχές όταν αδειοδότησαν αυτή τη μονάδα δεν, δεν υπήρχαν αλλαγές ή επεκτάσεις. Δεν ίσχυε λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η οδηγία αυτή. Όμως, το κύριο ζήτημα είναι αν η άδεια που δόθηκε το 2008 σε αυτή την μονάδα πληρεί τις προϋποθέσεις της ε, οδηγίας IPPC, της ε, ολοκληρωμένης δηλαδή οδηγίας για την καταπολέμηση της ρήπανσης. Ποιες είναι οι κύριες προϋποθέσεις εκεί και πάλι για τις υφιστάμενες μονάδες οι όροι της άδεια δυσφαλίζουν ότι ε, εκπληρώνονται οι κύριε υποχρεώσεις, δηλαδή ε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερες δυνατές ε, τεχνικές, θα πρέπει να αποφεύγεται η σημαντική ρήπανση και να υπάρχει και μηχανισμός παρακολούθησης. Ε, επίσης παρακολουθούμε το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Πρέπει λοιπόν να, γίνεται, ελέγχεται η ρήπανση από τα απόβλητα, η ρήπανση των υδάτων ή της ατμόσφαιρας που να προκαλείται από τη μονάδα. Αναλύθηκαν λοιπόν, αναλύθηκε η άδεια IPPC και έτσι κατάληξαμε το συμπέρασμα ότι ε, εκπληρώθηκαν αυτοί, αυτές οι προποθέσεις. Πράγματι, ε, εφαρμόστηκαν οι καλύτερε δυνατέ τεχνικές σε αυτή τη μονάδα. Υπήρξε έλεγχο ε, τη δραστηριότητα και του επίπεδου ρήπανση. Η άδεια στοχεύει στην αποφυγή της σημαντικής, ε, της μεγάλης ρήπανση. Υπάρχουν μέτρα για την αποφυγή της περιβαλλοντικής θαλάσσια ρήπανση. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για τον περιορισμό και τον έλεγχο της ρήπανσης που παράγεται από τις μονάδες αυτές υπάρχουν μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ατυχημάτων, είτε για να τα αποφύγουμε, είτε για να περιορίσουμε ε, τις επιπτώσεις των ατυχημάτων όταν αυτά ε, συμβαίνουν. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις είχαν εκπληρωθεί. Τώρα, αυτή η μονάδα έχει δύο μπόιλερ που ε, εκλείουν καπνούς και αέρια στην ατμόσφαιρα. Η άδεια επιβάλλουν ε, του ε, ελάχιστες ή μάλλον μέγιστες ε, τιμές για την ε, έκκληση διοξιδίου του άνθρακα, μονοξυδιού του άνθρακα και άλλων αερίων. Όλα αυτά πράγματι ίσχυαν όπως πρέπει. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του αέρα μέσα στη μονάδα και γύρω από τη μονάδα συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να ρυθμίσουμε ιδιαίτερη ρήπανση. Σύμφωνα με την άδεια υπάρχουν και αυστηρά ε, συστήματα παρακολούθησης για να ελέγχουμε τι εκλείται στην ατμόσφαιρα και αν αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για τη μείωση ε, των οσμών που εκλείονται από τις μονάδες έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα για την μείωση των οσμών ε, με τη χρήση θερ, διαδικασίας Τώρα για την θαλάσσια ρήπανση, για την ρήπανση των υδάτων, η οδηγία EPPC επιβάλλει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ε, έκκληση ε, μολυσμένων υδάτων στον υδροφόρο ορίζοντα. Υπήρχε ξεχωριστή ίδια μονάδα ε, διαχείρισης των υδάτων πριν από την απόρριψή του στον υδροφόρο ορίζοντα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η άδεια προβλέπει ότι όταν θα πρέπει να συμμορφώνεται αυτή η μονάδα ε, με το κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει να υπάρχουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα και προϋποθέσεις. Και πάλι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και λειτουργικό σύστημα. Επιπλέον, υπάρχουν μέτρα προστασίας ε, του εδάφους, ε, των υπογείων υδάτων, για τη διαχείριση ε, των υδάτων σύμφωνα, των αποβλήτων συγγνώμη, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Οι Ισπανικές αρχές επίσης μας ενημέρωσαν ότι έχουν διενεργηθεί επιθεωρήσεις στη συγκεκριμένη μονάδα και και υπήρξαν και πρόστιμα που επιβλήθηκαν ε, στους κατόχους. Οι επιθεωρήσεις αυτές έγιναν το 2010, τον Ιούνιο του 2010. Και εκεί είδαμε ότι ε, από την επιθεώρηση προέκυψε ότι σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία δεν ε, πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γι' αυτό και υπήρξε, οικονομικό, υπήρξε πρόστιμο. Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η άδεια που χορηγήθηκε σε αυτή τη μονάδα συνάδει με, τα, με τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και ιδιαίτερα με την οδηγία EPPC και όλες τις σχετικές οδηγίες, οδηγία περί ύδατος και ατμόσφαιρας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες ε, το ανώτερο δικαστήριο της Γαλλικίας ε, ακύρωσε τις άδειες που είχαν χορηγηθεί στη μονάδα λέγοντας ότι η άδεια αυτή δεν ε, συνάδει όχι με το κοινοτικό δίκαιο αλλά με τις εθνικές διατάξεις. Δηλαδή βρίσκεται πολύ κοντά σε οικιστικές περιοχές αυτή η μονάδα. Αλλά αυτό είναι εθνικό ζήτημα και έτσι έχει ακυρωθεί από το δικαστήριο η άδεια. Η περιφέρεια της Γαλλικίας έχει ασκήσει έφεση ε, στο αστικό δικαστήριο της Ισπανίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Εκτελεστική Επιτροπή για αυτές τις λεπτομερείς πληροφορίες. Η κυρία Άουκεν τώρα. Πολύ σύντομα από ότι κατάλαβα και σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Τα περισσότερα αυτά που άκουσα ήδη βρίσκονται στα έγγραφά μας. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, διότι έχω την εντύπωση ότι Είναι προβληματική η εγκατάσταση αυτή και μπορεί να, είναι, να πληρεί τους όρους της οδηγίας, αλλά Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να την κλείσουμε τώρα, με βάση την απάντηση που μόλις λάβαμε. Σας ευχαριστούμε. Και αν κανείς άλλος τώρα δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο, τότε μετά από όσα ακούσαμε θα ήθελα να προτείνω να παραμείνει ανοιχτό το θέμα της αναφοράς αυτής. Επίσης να διακόψουμε για ένα τεταρτάκι για μέχρι να ψηφίσουμε. Παρατέταρτο. Α, η κυρία Ναι, αφού έχουμε λίγο χρόνο και έχουμε τους ε, διερμηνείς, εγώ θα ε, θα ανέφερα το θέμα υπό τα διάφορα, αλλά θα το αναφέρω τώρα. Δεν είμαι ικανοποιημένη με τον τρόπο που επιβεβαιώνεται η μερίσια διάταξη. Τη λάβαμε σήμερα το πρωί. Είχαμε χθε την συνάντηση των συντονιστών. Και πιστεύω ότι η Πρόεδρος έκανε δραματική κατάχρηση του χρόνου μας. Χρησιμοποίησε όλο το απόγευμα για να στείλει ένα μήνυμα ουσιαστικά στην περιφέρειά της, ε, στην πατρίδα της, ε, που ε, δεν έχει πολύ σχέση με τη δουλειά μας. Νομίζω ότι μετά από αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια σωστή ημερήσια διάταξη που να συζητιέται και σωστά. Έχουμε τόσα πολλά θέματα, συχνά έχουμε τόση πίεση χρόνου Για παράδειγμα, κάποια θέματα έχουν αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη. Το θέμα του αερίου από σχιστόλιθο έχει αφαιρεθεί από το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να ε, μεταφέρουμε στην Πρόεδρο ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι, να λαμβάνουμε την ημερήσια διάταξη ε, μετά, το πρωί, μετά από τη συνάντηση των ε, συντονιστών, χωρίς χρόνο να το εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι η γραμματεία θα λάβει δεόντως υπόψη της, της παρατηρήσεις σας. Άρα λοιπόν για 15 λεπτά διάλειμμα.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 Σα ευχαριστώ πολύ.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 Καλημέρα, συνάδελφοι. Παρακαλώ, παρακαλώ στις θέσεις σας ε, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. I would ask you to... Παρακαλώ, μήπως μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε τις καρτούλες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Yeah. Are Έτοιμοι. Έτοιμες να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ ένας έλεγχος του συστήματος να δούμε αν λειτουργεί. Παρακαλώ συνάδελφοι, παρακαλώ συνάδελφοι, μπορείτε να ελέγξετε τις καρτούλες σας. Ξεκινάμε την ε, δίθεν ψηφοφορία. Ελέγχουμε λοιπόν να λειτουργεί το σύστημα. Ψήφισαν όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν πριν να ψηφίσουμε παρακαλώ την κυρία Βάλεαν, την εισηγήτριά μας, αν θα ήθελα να λάβει το λόγο. Καλημέρα συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και που προσπαθείτε να στηρίξετε την έκθεσή μου που δεν ε, ε, είναι για μας, ε, δεν είναι για τα κράτη-μέλη, είναι για τους πολίτες. Δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει το βασικό θεσμικό όργανο που υποστηρίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ό,τι έχω συμπεριλάβει στην έκθεση αυτά αναφερόταν λίγο πολύ στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Πολιτών. Προσπαθήσαμε να επικαιροποιήσουμε την έκθεση συμπεριλαμβάνοντας θέματα ε, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ε, αιτήματο ακόμα και μετά την ε, έκθεση της Κομισιόν. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να στηρίξουμε την έκθεση αυτή, το μήνυμα θα είναι ισχυρό προς τους πολίτες μας. Ιδιαίτερα σε αυτές τις μέρες αβεβαιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικού λόγους. Μπορούμε εμεί τουλάχιστον να δείξουμε ότι έχουμε μια κοινή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ένωσή μας. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους για τις τροπολογίες και τη δουλειά που έχετε κάνει με την έκθεση αυτή. Και κυρία Ματσόνη, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την εργασία σας. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία, παρακαλώ, για την έκθεση της κυρίας Βάλεαν για την ηθαγένεια της Ένωσης, όπως επίσης ότι θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε συμβαστική λύση 6. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. No, if it is necessary to check, yeah. Παρακαλούμε, αν θέλετε να το ελέγξουμε. Εντάξει, διαφορετικά συνεχίζουμε. Τροπολογία 54. Αποσύρθηκε. Συμβαστική λύση 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Φιλίπ Μπουλάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Χάνκης. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ακούγεται φωνή να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την τροπολογία 71 Χάνκης. Ηλεκτρονικά την 71. Πέρας τη ψηφοφορίας. Μισό λεπτό. Κάτι δεν λειτουργεί στην κυρία. Εντάξει, θα προσθέσουμε την ψήφο της συναδέλφου, αφού δεν λειτουργεί το μηχανήμα της. Εντάξει, ε, ναι, κατά είναι η κυρία Βίκστρομ και στο σύνολό της απορρίπτεται. 24 έως 25. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Η 73 Μπέκερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Κόζα Άγκης υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Και αν ψήφισαν όλοι. εγκρίνεται τελικά. 29, 11. 75 χάνκης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 πάξας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. συμβεστική λύση 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, κάτι να διευκρινίσουμε εδώ. Κάποιος ε, περισσεύει από τους φιλελεύθερους να ελέγξουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, η γραμματεία. ναι, σας καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά να ελέγξουμε. Μισό λεπτό.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 Παρακαλώ, παρακαλώ, οι συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες να κάνουν τον έλεγχό τους. Δηλαδή, είναι ακριβής ο αριθμός... Ε, ναι, η κυρία κάτι διορθώνει, οπότε μάλλον λύθηκε το πρόβλημα. Να προχωρήσουμε. 13, 13. 11. 11, 12, 13. Ακούγονται οι τρει αριθμοί. Παρακαλώ, κάθε ομάδα να επιτρέψει την ψηφοφορία μόνο από τον ε, σωστό αριθμό ψηφιζόντων. Παρακαλώ. Επόμενη ηλεκτρική ψηφοφορία. Και πάλι θα ελέγξουμε εκεί, εντάξει. Θα ελέγξουμε ποιοι ψηφίζουν από κάθε πολιτική ομάδα. Εντάξει, να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε παρακαλώ. Συμβιβαστική πρόταση 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ψηφίζουμε σε δύο χωριστά μέρη την παράγραφο 9. Το πρώτο μέρος της παραγράφου 9, η υπέρ του πρώτου μέρους της παραγράφου 9, κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε, παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παράγραφος 9, το πρώτο μέρος, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η κάρτα του κυρίου Μαρτίνες μάλλον δεν λειτουργεί. κ. Μαρτινές δείχνει ότι δεν λειτουργεί η κάρτα του, το σύστημα δηλαδή. Καταπίπτουν όλες οι επόμενες τροπολογίες. Πάμε στην παράγραφο 9, νέα. Τροπολογία 100. Αλφάνο Βάτιμα. Ξεχωριστή ψηφοφορία και πάλι. Πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα παράγραφος 10 νέα, 108 κόζα άγκης υπέρ, κατά, αποχές να ελέξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Δεν είδα και πολλά χέρια να ψηφίζουν. 108 κόζα άγκης. Άγκης, Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρα της ψηφοφορίες Μισό λεπτό να ψηφίσει και η κυρία Γκυγιόμ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κύριε Γκολόμ. Κύριε Γιγιόμ. Τι είστε υπέρ ή κατά. Υπέρ. Άρα λοιπόν προσθέτουμε μία θετική ψήφο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Αλφάνο βάτιμο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τροπολογία 109 αλφάνο βάτιμο ψηφίζουμε. Απορρίπτεται 14-14 το αποτέλεσμα. 110 Μπουλάντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κανονικά αλλά μισό λεπτό να κάνουμε και πάλι ένα έλεγχο ηλεκτρονικά ψηφίζουμε έλεγχος για την 114 και αν ψήφισαν όλοι Και πάλι 14-14. Ισοψηφία απορρίπτεται. 111 τροπολογία. Μότι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 μπάγκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 Κόζα Χάνκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 119 μπουλά υπέρ. 119. 119. Μπουλάν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ 119 μπουλάου ψηφίζουμε και αν ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 120 Ζανόκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. 125 μπουλάν υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν είδα καθαρά το αποτέλεσμα. 125 μπουλάν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Και αν ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 175 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 134 ψηφίζουμε παρακαλώ και αν ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 135 μπουλάν υπέρ κατά αποχές να αλλάξουμε και πάλι ηλεκτρονικά παρακαλώ 135 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας της ψηφοφορίας τροπολογία 136. Τι έγινε, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Να ψηφίσουμε και πάλι. Εντάξει. Ψηφίζουμε και πάλι Ψηφίζουμε και πάλι την 135 Μπουλάν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 135. Εγκρίνεται. 22-7 το αποτέλεσμα. Τροπολογία 100... Τροπολογία 136 Μπουλάν Λάρσκα Μπομπίνσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 137 Σντανόκα υπέρ κατά α, εγκρίνεται. Για την 139 προφορική τροπολογία κάποιος αντίθετος. Πώς είπατε. Κανείς δεν είναι αντίθετος με την ε, προφορική τροπολογία. Την 139 μετά από την τροποποίηση από την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 141 μπουλάν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142 μπουλάν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 μπουλά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 μπουλά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 τουργάις υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 η Τουργκάης υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 147 η Τουργκάης και αν ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 148. Ιτσεφ ε, Ιωτόβα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150. Νεντέλτσεβα. Σε δύο χωριστά μέρη. Καταπίπτει. Τι είπατε. Περνάμε στην 152. Ήλτσεφ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156. Μπουλάν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 157. Μπουλάν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158. Μπουλάν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 μπουλάν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμπαθητική πρόταση 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ...167 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 μπουλά υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ 168 μπουλά εγκρίνεται 169 μπουλά υπέρ κατά αποχές Να ελέξουμε και πάλι ηλεκτρονικά παρακαλώ. Δεν βλέπω τα χέρια σας. 169 μπουλά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 165. Μπουλά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται ήταν του κύριου Μπουλάου. 182 Μπουλάν και πάλι υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 183 Μπουλάν υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 184 Γκούσταυσον Γκουρμάη, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε παρακάτω για τις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1, μπουλά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, Γκούσταυσον Γκουρμάη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, μπουλά. Έχουμε προφορική τροπολογία τροπολογία. Κάποιος είναι αντίθετο με την ε, προφορική τροπολογία. Όχι. Άρα λοιπόν την ψηφίζουμε μετά την τροποποίηση από την τροπολογία. Την προφορική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Γκούσταυσον Γκουρμά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Σαλαβράκος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται επτά μπουλά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οκτώ μπουλά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εννέα κόζα χάνκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 του κυρίου Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική πρόταση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 μπουλά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 πάξας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 Βίλαντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 μπουλά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 δανόκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 μπουλά υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την 24 Μπουλάν. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 Μπουλάν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε για την 27 Μπουλάν. Πέρας ψηφοφορίας ηλεκτρονικής. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 28. Γκούσταυσον Γκουρμά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 30 μπουλάν υπέρ. Πώς είπατε? Ναι, ταυτόσημη. Τότε η 32, Γκούσταυσον Γκουρμάη, υπέρ της 32, κατά αποχές απορρίπτεται. 34, Μπουλάν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35, Μπουλάν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος ε, λατινικό H. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Κα... Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει, ελέγχουμε. Για το H το λατινικό. Πέρα της ψηφοφορίας της ηλεκτρονικής. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 Πάξας Πώς είπατε? Όχι, όχι. Καταπίπτει. Πάμε στην συμβαστική πρόταση 3. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. 42 είπαμε. 42 μπουλά υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Δεν βλέπουμε τι υπερίσχυσε. Το 42 λοιπόν, 42 τροπολογία Μπουλάμ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 43 Χάνκις. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «44». Μόνο το δεύτερο μέρος ψηφίζουμε. Καταπίπτει το πρώτο μέρος, γιατί η 45 εγκρίνθηκε. Όχι, όχι. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, ψηφίζουμε τη 45, Βίλαντ, υπέρ, κατά, απόχες να ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά για τις 45 Βίλαντ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 45. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται 44 σε χωριστά μέρη, μόνο το δεύτερο μέρος για το πρώτο καταπίπτει. Δεύτερο μέρος, υπέρ παρακαλώ, δεύτερο μέρος 44, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβατική πρόταση 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία Ψηφίζουμε επί του συνόλου. Πέρας ψηφοφορίας. Τι έγινε. Εντάξει. Εγκρίνεται. 24-1. Κυρία Βάλεαν, συγχαρτήρια για την έγκριση αυτή. mais toi, tu as particulièrement

Doamnelor și domnilor, vă rog frumos puțină liniște. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, λίγη ησυχία. I'll ask you to be quiet, please. Παρακαλώ, ησυχία, ησυχία. Φτάσαμε στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η 354 του 2006 αναφορά Rodney Mail Βρετανικής Ιθαγένειας σχετικά με ρήπανση της δημοθάλασσας του Κλέντο ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των δύο εταιριών Exxon και Quater. Ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στον Rodney Mail, στον κύριο Rodney Mail, αναφέροντα. Παρακαλώ. Το λόγο έχει ο κύριος Rodney Mail αναφέρον. Παρόν ο κύριος Είναι παρόν ο κύριος Παρακαλώ. Rodney Μέιλ, Είναι ο αναφέρον. Ποιο ήταν το ερώτημά σας, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βιομηχανία υγροποιημένου αερίου γνωρίζουν ότι υπάρχουν διαρροές ε, στις δεξαμενές. Γι' αυτό γιατί απλώς παρακολουθεί η βιομηχανία όταν η λιμνοθάλασσα συγκεκριμένα επελέγει ω τόπος που έπρεπε να ε, μπουν και να παραμείνουν ε, τέτοιες δεξαμενές. Προ, προφανώς και πρόκειται για μεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον και για τους κατοίκους. Όμως γιατί η βιομηχανία δεν ανέφερε ότι είναι το τελευταίο και χειρότερο λιμάνι που θα έπρεπε να επιλεγεί και θα έπρεπε να απαγορευτεί η είσοδος ε, σε τέτοια σκάφη και για το, ε, και για το φορτίο αλλά και για το προσωπικό, το πλήρωμα που αυτή τη στιγμή ε, 15.000 προσωπικού που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν ε, σε περίπτωση ατυχήματος. Σύμφωνα με έρευνες ανακαλύφθηκε ότι το, το Σεπτέμβριο του 2011 υπήρχε σημαντική διαρροή θα μπορούσε αυτό να έχει οδηγήσει σε οδυνηρές συνέπειες. Αυτό το συζήτησα με τους πολίτες του Waterstone και αν όχι γιατί όχι. Ε, τι αυτό θα σημαίνει, τι θα σήμαινε μια πυρκαγιά για παράδειγμα για τους ε, κατοίκους ε, του, της ε, περιοχής. Ε, σε αντίστοιχη περίπτωση στην Αριζόνα και στη Γαλλία είδαμε ότι υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Αυτό θα οδηγούσε και σε πυρκαγιά στην άλλη δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου ή θα οδηγούσε πυρκαγιά σε ε, άλλα είδη καυσίμων που ήταν αποθηκευμένα δίπλα εκεί πόσες ζημιές θα είχαν προκληθεί και πόσες, ε, πόσοι θάνατοι θα είχαν προκληθεί από όλο αυτό το ε, συμβάν. Ας το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες. Ήταν σωστό να επιτρέψουμε να υπάρχουν τέτοιες δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου δίπλα στις υπόλοιπες δεξαμενές. θα πρέπει να επαναξετάσουμε ε, την λειτουργία τέτοιων ε, χώρων γιατί το να φέρουμε τέτοια φορτία LNG ε, σε, σε τόσο μικρούς λιμένες με μικρό περιθώριο λιγμών και με βράχους αυτό σημαίνει ότι με ένα πολύ μικρό ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο έως και 50.000 ανθρώπους. Το φορτίο δεν είναι, το σκάφος δεν είναι δύσκολο, το, συγγνώμη, το σκάφος δεν είναι επικίνδυνο, το φορτίο του είναι επικίνδυνο. Αυτό καθιστά και το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο επικίνδυνο, γιατί είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο ε, αέριο και, το οποίο είναι σε υγρή μορφή, σε, μια, σε 53 βαθμούς, αν πάει στο μείων 162 γίνεται και πάλι αέριο. Γι' αυτό όταν βγαίνει από την δεξαμενή, ε, επιστρέφει σε μορφή αερίου με όγκο 600 φορές μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναμειχθεί με τον αέρα ε, πριν υπάρχει ανάφλεξη. Εγώ θα ήθελα πριν δοθεί άδεια να ε, μπει τέτοιο σκάφος στο λιμένα, θα πρέπει να υπάρχει ένα πιστοποιητικό ασφαλείας. Αν αυτό λειτουργούσε πριν από το 2003, οι αρχές θα είχαν έρθει αντιμέτωπες με όλες αυτές ε, τις ερωτήσεις που δεν απάντησαν όταν έλαβαν την ε, απόφαση ο λιμένας έχει σχεδιαστεί για να ε, προστατεύει τους κατοίκους και τους εργαζομένους. Δόθηκε άμεση απόφαση, αλλά αυτό δεν ε, διασφαλίζει την ασφάλεια των ε, κατοίκων και των εργαζομένων. Και τώρα έχουμε 50.000 κατοίκους που μένουν δίπλα σε αυτή τη λιμνοθάλασσα και βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο από εγκάβματα ή ακόμα και από τέφρωση πρέπει να παραμείνουμε στις βέλτιστες πρακτικές, δηλαδή σε έναν άριστης ποιότητας λιμένα που θα αποφεύγει τους κινδύνους. Και εκεί θα δείτε ότι η συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα απέχει τόσο πολύ από τα καλύτερα πρότυπα για ένα λιμένα που ε, αν επιτρέψουμε αυτή την κατάσταση, τη συνέχιση της κατάστασης, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την απειλή θανάτου που ε, ε, κρεμάται πάνω από τα κεφάλια όλων αυτών των κατοίκων που κινδυνεύουν από ένα ενδεχόμενο ατύχημα και από ένα κίνδυνο που μπορεί να αποφευχθεί και δεν απεφεύχθη γιατί οι αρχές ε, αποφάσισαν να, να παραβλέψουν τις βέλτιστες πρακτικές και δεν δημιούργησαν έναν καλής ποιότητας λιμένα που θα έπρεπε να απαγορέψουν την αποθήκευση τέτοιου αερίου ε, σε απόσταση τριών μιλίων από τις ε, κατοικούμενες περιοχές. Λόγω αυτών των τεράστιων κινδύνων, αν υπάρχει κάποια διαρροή, αυτό βάζει σε άμεσο κίνδυνο ε, τους κατοίκους, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ασφαλές σημείο για τους κατοίκους στα επόμενα πέντε μίλια ούτε μεγάλο περιθώριο ελιγμού ε, των ε, σκαφών μέσα στο λιμένα. Είναι λοιπόν επικίνδυνο λιμάνι. Ε, οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει μέσα σκάφος με LNG και αυτό θέτει σε κίνδυνο και τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κοντά σε αυτή την περιοχή. Άρα, το βρήκα. Πρέπει να θυμούμαστε ότι εφόσον αυτές οι αρχές δεν ε, ε, εφαρμόζουν τις ε, κατάλληλες οδηγίες και όλα αυτά για λόγους κόστους, για να μην επιβαρύνουν τον προπολογισμό αυτών των project, αυτών των σχεδίων. Και έτσι αγνόησαν τους κινδύνους και τις απειλές. Οι δεξαμενέ αυτές λοιπόν είναι επικίνδυνες και καμία αρχή δεν έχει παρέμβει για να αποσοβήσει αυτόν τον κίνδυνο. Η Πρόεδρος διακόπτη. Συγγνώμη, πρέπει να σας ε, ζητήσω να διαβάζετε λίγο πιο αργά, γιατί δεν σας παρακολουθούν οι διερμηνείς. Ο γιατρός Τόνι Κόξ, ειδικό στα θέματα, αναφέρει ότι ε, δεν έχει γίνει η απαραίτητη αξιολόγηση αντικτύπου για τους κατοίκους. Και γιατί έγινε αυτό. Η μη διεξαγωγή αυτής, αυτής της αξιολόγησης αντικτύπου σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τους κινδύνους ε, για τους κατοίκους και, σε αυτό σημαίνει ότι αυτός ο λιμένος δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ποτέ για, ε, τα, για τις δεξαμενές και αυτά τα σκάφη αν ακολουθούσαμε τις βέλτιστες πρακτικές για αυτό το λιμένα, τότε δεν θα λάμβανε ο λιμένας το πιστοποιητικό ασφαλείας, γιατί είναι πάρα πολύ οι ε, κίνδυνοι. Και έτσι δεν θα πληρούσε τα κριτήρια ασφαλείας. Γι' αυτό θα έπρεπε να επανεξετάσουμε το πιστοποιητικό ασφάλειας και, για να, και να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους για να δούμε πόσοι κάτοικοι κινδυνεύουν για όλα αυτά τα λιμάνια που δεν πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφαλείας. Δεν έχει γίνει εξολόγηση αντικτύπου ε, σε καμία αποβάθρα ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περίπτωση πυρκαγιάς στο λιμένα είτε σε ε, σκάφος που βρίσκεται εν πλώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει ποτέ δυνατότητα χρήσης ε, αυτού του λιμένα από σκάφη με υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες. Για παράδειγμα, αν βυθιστεί ένα τέτοιο σκάφος στο λιμένα, λέτε ότι είναι αδύνατο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Και υπάρχουν και άλλα σενάρια που μπορούν να φανταστεί κάποιο ως χειρότερα σενάρια. Πάντα εξαρτάται το τι θέλουμε να συζητήσουμε. Αν βυθιστεί λοιπόν ένα τέτοιο σκάφος, μπορεί να ε, μπορεί να γύρει και να οδηγήσει στη διαρροή ε, εκατομμυρίων τόνων φυσικού αερίου. Και έτσι η μετάβαση από το φυσικό αέριο, από το LNG σε μεθάνιο ξεκινά και έτσι το LNG γίνεται και πάλι ε, μετατρέπεται σε αέριο με, με όγκο 600 φορές μεγαλύτερο. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν ε, τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό βεβαίως ε, και θα κατέστρεφε ολόκληρο το λιμένα. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο που μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό δεν είναι δυνατόν σε έναν ε, λιμένα που ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές. Αλλά φανταστείτε, σε ένα τέτοιο σενάριο, ολόκληρος ο λιμένας βυθίζεται ε, σε μεθάνιο και πάλι σε θερμοκρασία μείον 160 ε, βαθμών Κελσίου. Γιατί είναι πολύ πυκνό, πολύ κρύο, βαρύτερο από τον αέρα, ε, κινείται γρήγορα, διαχέεται γρήγορα. Δεν θα υπάρχει ανάφλεξη εκεί γιατί πρέπει να ανακατευθεί, να αναμειχθεί 10 ακόμα φορές με την ατμόσφαιρα για να έχει, υπάρχει σωστή αναλογία μεθανίου και αέρα. Το μεθάνιο βεβαίως και είναι θανατηφόρο σε τέτοια συμπίκνωση για τον άνθρωπο. Και βεβαίω φανταστείτε τι γίνεται μετά όταν υπάρχει ανάφλεξη και έχουμε θερμοκρασίες χιλίων και 2.000 βαθμών Κελσίου. Μια τέτοια καταστροφή λοιπόν ε, θα μπορούσε αντιστοιχεί σε 45 ε, βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χειροσύμα. Επομένως, αν υπήρχε ένα τέτοιο πιστοποιητικό ασφαλείας, θα έπρεπε να έχει δοθεί μόνο από την αρμόδια αρχή και να διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση αυτή συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές. Τότε δεν θα είχε δοθεί άδεια για τον ελιμενισμό τέτοιων σκαφών, γιατί ήταν προφανές ότι ε, επέσυρε κίνδυνο θανάτου για του 50.000 κατοίκου τη ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και δεν θα είχε δοθεί άδεια. Θα είχε απορριφθεί το αίτημα κατασκευή ε, τέτοιου λιμένα και θα είχε μεταφερθεί ο λιμένα αλλού, σε κάποιο άλλο ασφαλέστερο σημείο στον Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει λοιπόν ασφαλής περιοχή ε, που αποκλείει τις ε, πηγές ανάφλεξης και θα έπρεπε να υπάρχει ένα, ε, ένα εμπόδιο 2-5 μιλίων για την ασφάλεια των κατοίκων, γιατί σε περίπτωση ανάφλεξης μέχρι εκεί πάει το αέριο. Γι' αυτό μέχρι να εξακριβωθεί με ελέγχους και μέχρι να γίνουν όλα αυτά μάλλον μέσω ελέγχου, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το, αυτή η ζώνη αναχέτηση των 2-5 μιλίων. Όλοι στην περιοχή ξέρουν ότι δεν ακολουθούνται βέλτιστες πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας επικίνδυνος λιμένας, ιδιαίτερα για όσους μένουν ε, εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αγνοούν λοιπόν τους κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Δεν είναι κατάλληλος ε, ο λιμένας αυτός. Πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος και για τα πληρώματα των σκαφών και για τους κατοίκους. Πρέπει να απαγορευτεί λοιπόν ο ελιμενισμός σκαφών με υγροποιημένο αέριο. Επειδή ήδη λειτουργεί αυτός ο λιμένας με πηγές ανάφλεξης παντού, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους κατοίκους που μένουν κοντά στη λιμνοθάλασσα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να επιτρεπεί η είσοδο στο λιμένα για τέτοια σκάφη. Γιατί αν υπάρξει ένα συμβάν, ένα ατύχημα, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια ε, για τους 50.000 κατοίκους. Το καταστροφικό φορτίο ε, των σκαφών αυτών θα οδηγήσει σε τεράστιες ζημιές και θανάτους. Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν. εάν οικοδομηθεί ένας νέος λιμένας. Right. Um, there are number of other points, of course. Υπάρχουν βεβαίω και άλλα σημεία. Το σχέδιο της ανάγκη, το οποίο δεν ε, επιτρέπεται να συζητηθεί μέχρι την οικοδόμηση, η κατασκευή αυτών των δεξαμενών, θα έπρεπε να συζητηθεί στην αρχή Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγερ, για την ε, παρουσίασή σας. Ήταν μακροσκελής, όμως, γι' αυτό θα ε, ζητήσω από τους άλλους αναφέροντες να είναι πιο σύντομοι. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρίσος Μπάξτεν. Ε, good morning. Thank you, Madam Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Είμαι ε, δικηγόρος της Safe Haven, ε, της Οργάνωσης ασφαλου, ε, του Ασφαλιλούς Λιμένα και έχω διανύμει κάποια έγγραφα τα οποία ελπίζω ότι θα σας είναι χρήσιμα και το 2007 παραπονεθήκαμε για την ίδια υπόθεση και μετά. Ε, τα βασικά μου σημεία είναι τα εξής. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να περιμένουν από τις ε, κυβερνήσεις τους ε, να τηρούν τον νόμο. Αυτό δεν έχει γίνει στην περίπτωση αυτή. Οι δημόσιες σχέσεις δεν αρκούν. Είμαστε ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά τους και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας βοηθάτε με αυτό το πολύ δύσκολο θέμα. Ε, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, μπορώ να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ε, του πώς ε, ε, προχωράνε τα πράγματα. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η θαλάσσια πτυχή των λιμένων για υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι η πιο επικίνδυνη πτυχή. Λείπουν ε, αξιολογήσεις κινδύνου και από ό,τι βλέπουμε δεν έχουν εκπονηθεί αυτές οι μελέτες. Και σύμφωνα με την οδηγία ε, για τις μελέτες περιβαλλοντικού τεκτύπου έπρεπε να έχουν γίνει αυτές οι μελέτες. Έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λάβαμε απόφαση από ε, ε, ένα από τα σώματα του δικαστηρίου που λένε ότι παρότι ήταν, ε, υποβλήθηκε πολύ σωστά η προσφυγή αυτή, η κυβέρνηση έκανε αρκετά διότι είχε παράσχει ένα σωρό πληροφορίες. Η παροχή πληροφοριών οι πληροφορίες αυτές όμως δεν ε, εξετάστηκαν. Ε, αυτό το ανέφερε και ε, ο κύριος Μέιν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι πληροφορίες ότι δεν αρκεί να παρέχει κανείς απλά πληροφορίες στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων. Θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου. Και ε, με αυτό ακριβώς θέλουμε να προσφύγουμε ε, στο, σε ανώτερο επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρκεί δηλαδή για τις κυβερνήσεις απλά να παρέχουν πληροφορίες ε, για να μην πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις. Και ε, γι' αυτό ακριβώς είναι κρίσιμη η δράση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Ε, είναι σαφές ότι οι ε, περιβαλλοντικές δηλώσεις ήταν λυπείς όσον αφορά την ασφάλεια και τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ε, έχουν πιέσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για πληροφορίες, αλλά από ό,τι καταλάβαμε δεν έχουν δοθεί οι πληροφορίες αυτές. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσετε να ε, πιέζετε την κυβέρνηση και ενδεχομένως να ξεκινήσετε διαδικασία παράβασης. Αυτά θέλω να πω και να προσθέσω ένα ακόμα πράγμα κυρία Πρόεδρε. Στο χαρτί που σας έχω μοιράσει συμπεριλαμβάνεται αυτό. Μπορεί να μην το βλέπετε καλά, σας δείχνω όμως το χαρτί αυτό. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το χαρτί αυτό, διότι δεν περιέχει καμία πληροφορία. Πρόκειται για πληροφορίες για ένα σχέδιο άμεσου δράσης ε, το οποίο υποτίθεται ότι είναι, ε, είναι διαθέσιμο στο κοινό. Έχουν διαγραφεί όμως ε, τα στοιχεία σύμφωνα με, τον, με τους κανόνες για τις ε, προσβάσεις στα έγγραφα. Ε, μόνο οι μόνες λέξεις που ε, φαίνονται στο έγγραφο αυτό είναι ε, το νέφος ε, εξαρμίσεων που μπορεί να δημιουργηθεί. και αυτό ανέφερε και ο προλαλή σα. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να μα βοηθάει στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σα. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Μπράκεν από του αναφέροντε. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, κύριε Βαπράκεν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Οι δύο προλαλήσαντες κάλυψαν πολύ καλά το θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σας σε μια πρόσφατη εξέλιξη στον Λιμένα. Ακούσατε ε, για την διαρροή σε, έναν από, σε μια από τις εξαμενές στο Waterstone. Πριν ε, ξεκινήσει η κατασκευή, μας ε, ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση διαρροής. Όταν λοιπόν η ομάδα μας άκουσε ε, κάποιες φήμες για διαρροή, ε, ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία και ο και η Υπηρεσία υγεία και Ασφάλειας ε, που είναι η αρχή που είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών στο κοινό για θέματα υγείας και ασφαλείας και φυσικά και για τη ρύθμιση των ε, προϋποθέσεων για ασφαλείας και υγείας στις ε, σχετικές εταιρείες μας είπαν ότι πράγματι υπήρξε μια μικρή διαρροή. Αυτό έγινε ήδη τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε Ε, έχω ζητήσει πληροφορίες από την υπηρεσία αυτή και φαίνεται σαν να υπάρχει μια ανατροπία μυστικότητας γύρω από το θέμα αυτό, διότι ακόμα και τώρα η αρχή αυτή αρνείται να καθησυχάσει την κοινότητά μας ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι διαρροές. Δεν μπορούν καν να μας πούν αν συνεχίζει να υπάρχει διαρροή. Νομίζω ότι οποιοδήποτε στην αίθουσα ετούτη, αν αντιμετώπισε την κατάσταση αυτή, ε, θα έφρυτε με την κατάσταση και θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι επιπλέον η λιμενική αρχή με το θράσος που έχει αποκτήσει επειδή μπόρεσε ε, να παρακάμψει τόσους από τους κανόνες που υποτίθεται ότι θα πρέπει να τηρεί, ανακοίνωσε νέα κατασκευή ε, στον Λιμένα, όπου θα, ε, ε, όπου θα φτάνουν κρουαζιερόπλια. Τώρα λοιπόν θα αρχίσουν τα κρουαζιερόπλια να μπαίνουν στο λιμάνι Milford Haven και πιστέψτε το, αυτά τα κρουαζιερόπλια θα βρίσκονται ακριβώς δίπλα ε, στα πλοία ε, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Όχι μόνο θα βρίσκονται δίπλα στα πλοία αυτά, αλλά θα βρίσκονται και στο πιο στενό μέρος του, της διαδρομής ε, που θα πρέπει να περνούν τα πλοία με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Εγώ το μόνο που ζητώ από την Επιτροπή σας είναι να προσπαθήσει ε, να πιέσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ε, πληρεί την υποχρέωσή της απέναντι στους πολίτες ε, για ασφάλεια και υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε πώς έχει κατάσταση. Και τώρα η κυρία Ζίμπελ ε, θα λάβει το λόγο πάλι για να μας ε, πει μερικά πράγματα για την υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Το βασικό ζήτημα της ε, Επιτροπής κατά την εξάρτηση αυτής της αναφοράς ήταν ο ισχυρισμός ότι οι θαλάσσιοι κίνδυνοι δεν αξιολογήθηκαν σε αυτό το συγκεκριμένο λιμάνι και ακόμα κι αν είχαν αξιολογηθεί δεν δόθηκαν αυτά τα στοιχεία στην δημοσιότητα και σίγουρα όχι στους αναφέροντες. Δεν θέλω να πω τα όσα έχουμε ήδη παρουσιάσει, τα οποία έχετε στη διάθεσή σας, αλλά ήδη από το Μάιο του 2007 στην οδηγία Σερβέιζα ε, για τον έλεγχο μεγάλων κινδύνων από επικίνδυνες ε, ουσίες δεν ισχύει εδώ. Οι ουσίες που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής ναυσιπλοείας ε, δεν ισχύει εδώ πέρα. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό, το, αυτή η νομική πράξη, παρόλο που η Σεβέζο 2 αναθεωρείται αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στην ε, διαδικασία πρώτης ανάγνωσης. Όσο έχει τώρα η κατάσταση και όσο είχε για τη ε, φάση αδειοδότησης του προγράμματος, η Σεβέζα 2 δεν ε, ίσχυε για τους θαλάσσιους κινδύνους. Υπάρχει και μία άλλη οδηγία περιβαλλον... αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διεξήχθη και εκεί υπήρχε και ενημέρωση του, της κοινή γνώμης. Και αυτό ανέφερε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερα σε μια συνεδρίαση όπως συναντήσαμε του αξιωματούχου του Ηνωμένου Βασίλειου του 2010 και εκεί είπαμε ότι κατά την Επιτροπή θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί οι θαλάσσιοι κίνδυνοι υπό την ε, οδηγία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διαφώνησε και καταλήξαμε σε μια πρακτική λύση. Δηλαδή συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε και ζητήσαμε από τον Ηνωμένο Βασίλειο να δώσει σε εμά και στην κοινή γνώμη ε, πληροφορίε και στοιχεία που είχαν ε, για, τη, για τους θαλάσσιους κινδύνους. Ανέλαβαν λοιπόν το καθήκον να ε, δημοσιεύσουν αυτές τις πληροφορίες μέσω χαρτών, δηλαδή με μια μορφή χάρτη με επιπρόσθετες πληροφορίες και μας είπαν ότι θα το έκαναν αυτό μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Πέρασε αυτή η προθεσμία, δεν λάβαμε τις ε, πληροφορίες αυτές και έτσι ξεκινήσαμε ένα, αυτό που ονομάζουμε EU Pilot, δηλαδή ένα επίσημο αίτημα προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να μας παράσχει τις ε, απαιτούμενες πληροφορίες. Συναντηθήκαμε με αυτές τις αρχές στα τέλη Ιανουαρίου και μας είπαν ότι πράγματι υπάρχει καθυστέρηση και ότι η νέα προθεσμία θα είναι ο Ιούνιος του 2012. Προφανώς και πρόκειται για σημαντική καθυστέρηση. Μόλις λάβαμε την επίσημη ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα θα δούμε αν θα κινήσουμε διαδικασία επί παραβάση υπό το άρθρο 258 της συνθήκης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα μας είπατε και παρακαλώ η συνάδελφος Evans Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους ε, αναφέροντες ε, στην Επιτροπή μας σήμερα. Η αναφορά θεωρήθηκε παραδεκτή τον, ε, Δεκέμβριο του 2000, τον Σεπτέμβριο του 2006. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί το καιρό. είμαι ευγνώμων προς την Επιτροπή για όλη τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό, διότι Ε, είναι προφανές ε, το επίπεδο ε, ενδιαφέροντος που υπάρχει για το θέμα αυτό και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το Δέλτα του Ποτάμου Κλωτέη στην Ουαλία, στην περιφέρειά μου τους, τους ανθρώπους εκπροσωπώ εγώ και ε, φυσικά υπάρχει σημαντική απειλή για την υγεία των ανθρώπων και για τις περιουσίες τους και στην ε, περίπτωση αυτή η Κομισιόν όπως είπε θεωρεί ότι οι ε, αρχές της, ε, του, ε, του, του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν παραβιάσει την νομοθεσία. Θα έπρεπε το θέμα αυτό να ε, έχει καλυφθεί ε, στα πλαίσια της αρχικής ε, μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου. Έχουμε ακούσει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το αμφισβητεί αυτό και υπήρχε η συμφωνία αντί να προσφύγει η Κομισιόν κατά του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει τους χάρτες, ε, τις πληροφορίες ε, που ήδη υπήρχαν όσον αφορά ε, τις διαδικασίες ασφαλείας και ότι όλες οι πληροφορίες αυτές θα, έπαιρναν, θα έμπαιναν στον απαραίτητο μορφότυπο και θα θα ήταν έτοιμες μέχρι τον προηγούμενο Οκτώβριο. Αυτό δεν έχει συμβεί. Ακούσαμε όλες ε, τις ανησυχίες. Ε, ακούσαμε και για τη διαρροή πέρσι τον Οκτώβριο. Ε, έχει διανεμηθεί επιστολή σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας σχετικά με το θέμα αυτό. Το... Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όμως αρνείται να δεχθεί ότι δεν έχει τηρήσει την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μελέτη αντικτύπου και την αξιολόγηση κινδύνων. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό θέμα ε, όσον αφορά την ερμηνεία αυτή τη οδηγία από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν ε, σημαντικά θέματα όσον αφορά την, ε, το δικαίωμα πληροφοριών. Είδαμε αυτό το γελίο έγγραφο που έχουν διαγραφεί όλε οι απαραίτητες πληροφορίες όταν οι κάτοικοι ζήτησαν σχετικέ πληροφορίε. Και στο μεταξύ, οι, οι ντόπιοι στο Milford Haven δεν γνωρίζουν τι μέτρα έχουν ληφθεί για να προστατευτεί η υγεία τους ε, και να προστατευτούν οι κατοικίες τους και συνεχίζουν να ανησυχούν. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η άμεση δράση για να ε, αποκατασταθεί η κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ πάνω στο θέμα αυτό και προτείνει ε, να ε, καθυστερήσει μέχρι τον Ιούνιο, τη στιγμή που είπαν ότι ε, οι, πληροφορίες, οι απαραίτητες πληροφορίες όλες υπάρχουν, απλά θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε την κατάσταση και παρακαλώ την Επιτροπή να σκεφτεί το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης, να μην δεχτεί αυτή την προθεσμία και να ασκήσει πραγματική πίεση στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι ο κόσμος θέλει να γνωρίζει ότι είναι ασφαλής. Εάν δεν έχουμε τις πληροφορίες αυτές, ε, ο κόσμος ε, θα ζει με φόβο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Ελμέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μέιλ για την ιδιαίτερα μακροσκελή, επαναληπτική και μελοδραματική παρουσίαση Ομολογώ ότι όταν ε, τα άκουσα όλα αυτά, ε, ε, η αντίδρασή μου ήταν ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αιμονή με την ασφάλεια και την υγεία και ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει καν να τα εξετάσουμε. Αλλά από τα όσα άκουσα μετά από αυτό πρέπει να πω επίσης ότι εξεπλάγει που η Βρετανική κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει αυτές τις πληροφορίες και πράγματι οι κάτοικοι καλά κάνουν και ανησυχούν και δικαιούνται κάποια στοιχεία, μια ενημέρωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει η Βρετανική κυβέρνηση να παράσει αυτές τις πληροφορίες και πράγματι η Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσει πιέσει στην Βρετανική κυβέρνηση για να ενημερώσει τους κατοίκους τα όσα ακούσαμε στο τέλος της συζήτησης πραγματικά δημιουργούν ανησυχίες και θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν οι πληροφορίες. Τι αξιολόγηση αντικτύπου έχει γίνει, ποιο είναι το σχέδιο έκτακτη ανάγκης και ποια είναι τα επίπεδα επικινδυνότητας. Ο κύριος Μέιλ νομίζω δεν, δεν τις μέτρησε, αλλά νομίζω ότι έκανε 30-40 ερωτήσεις. Οι περισσότερες από αυτές ήταν τεχνικής ε, φύσεως. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό όσοι πράγματι είναι αρμόδιοι να απαντήσουν, να το κάνουν. Thank you for your on of the... Ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση. Τώρα θα δώσω το λόγο σε έναν από τους ε, τρεις ε, αναφέροντες. If you have something to add, the petitioners. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε. but very briefly. But very briefly, please. Thank you. Um, Πολύ σύντομα, μας παρακαλώ. Μάλιστα. Ένα από τα προβλήματα που εντοπίζω, πέρα από τα 35 διαφορετικά σενάρια μπορεί κάποιος να σκεφτεί, είναι το εξής. Αν βυθιστεί ένα τέτοιο σκάφος στο λιμάνι, μάλλον αν ένα ε, συμβατικό πλοίο ε, με πετρέλαιο βυθιστεί, τότε μόνο το, το πετρέλαιο θα, θα διαχυθεί στην ε, θάλασσα. Ενώ η διαφορά με το φυσικό αέριο είναι ότι θα σκοτώσει και του 50.000 κατοίκους τη ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η διαφορά. Σα ευχαριστούμε προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις όλες εξελίξεις. Το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το 17. Μισό λεπτό. Ε, Συνεχίζοντας λοιπόν, θα παραμείνει ανοιχτό το θέμα της προηγούμενης αναφόρας για τη ρήπανση αυτή και στις αρμόδιες αρχές για την υγεία και την ασφάλεια θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους και επίσης θα έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για διευκρινήσεις. Όπως επίσης θα έρθουμε σε επαφή ξανά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε στην ημερήσια διάταξη 17 σχετικά με το πόσιμο νερό με την προσθήκη φθοριοπυρητικού οξέως 2010-2007 του Ρόμπερτ Πόκοκ εξονόμαστε της οργάνωσης Voice of Irish Concern for the Environment και η δεύτερη 210 του 2007 του Walter Graham Βρετανικής Ιθαγένειας εξ ονόματος του Συμβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας κατά της ε, φθορίωσης. Παρακαλώ, κ. Πόκοκ. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που επιμένετε ε, στην αναφορά αυτή για την ε, φθορίωση του νερού διότι πολλοί κάτοικοι ε, της ε, Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ε, το τόπο τελευταία ίστα της προσφυγής ε, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτή την πολιτική. Θα ήθελα να καλύψω το θέμα από τρεις πλευρές. Καταρχήν να σας θυμίσω ποια ήταν η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλές ερωτήσεις ευρωβουλευτών τα τελευταία χρόνια. Ήταν να ληφθεί γνωμοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή για τους ε, κινδύνους προς την υγεία και το περιβάλλον. Να ε, σας συνοψίσω την ανάλυση που μας έδωσαν. Και θα ήθελα να απευθυνθώ πάλι στην Επιτροπή και να πω ότι η απάντηση που λάβαμε στο θέμα αυτό ε, ήταν τελείως ανεπαρκής ε, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Η αναφορά αυτή, ε, τελευταία φορά που υπολήθηκε στην Επιτροπή ήταν τον Μάιο του 2008 που φαίνεται σαν να είναι πολύ καιρό οι ευρωβουλευτές ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προ το τέλο ε, τη χρονιά αυτή, λοιπόν, ε, παρενέβη και ζήτησε αξιολόγηση κινδύνου από την Επιστημονική Επιτροπή ε, για κινδύνου προ την υγεία και, και το περιβάλλον, την ΣΕΡ. Η προκαταρθική γνωμοδότηση το, δημοσιεύτηκε το 2009 και επιβεβαίωσε την ε, μη διακριτική φύση αυτής της, ε, της ε, φαρμακευτικής αγωγής. Θεώρησε ότι η φθορίωση του νερού αποτελεί ένα πολύ χοντροκομμένο μέσο χωρίς ε, να υπάρχει σαφές κατόφλι. Ε, είναι σαφές αυτό, πρόκειται για φαρμακευτική αγωγή και οδηγεί σε ζημιά. Η Επιτροπή ΣΕΡ, λοιπόν, ε, οργάνωσε δημόσια ακρόαση με τους ενδιαφερομένους το Σεπτέμβριο του 2010 εδώ στις Βρυξέλλες. Και να σας πω κάτι σχετικά με τη συγκεκριμένη αυτή δημόσια ακρόαση. ήταν πολύ ευχάριστο για οποιονδήποτε από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ή οποιονδήποτε που ενδιαφερόταν για αυτήν την πολιτική, διότι για πρώτη φορά έγινε ανοιχτή ειλικρινή ε, συζήτηση. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ε, ε, απήντησαν ε, με πολύ σωστό τρόπο στα ερωτήματά μας. Μια τέτοια συνάντηση θα ήταν αδύνατο να γίνει στην Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά την πολιτική φθορίωση, υπάρχει ένα νέφος καπνού το οποίο έχει οργανωθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Α επανέλθουμε λοιπόν τώρα στη γνωμοδότηση της ΣΕΡ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2009, πριν σχεδόν δύο χρόνια. Δεν, ε, έχει υιοθετηθεί, ε, δεν έχουν υιοθετηθεί συμπεράσματα ούτε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε τη Ιρλανδία. Ε, το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται φθορίωση για την κανονική του ανάπτυξη στην Ιρλανδία ε, μας λένε τακτικά ότι όλοι πρέπει να λαμβάνουν και μάλιστα μέσω του νερού που δεν μπορούν να το αποφύγουν. Η ΣΕΡ επίσης ε, κατέληξε ότι η ε, υπερβολική λήψη φθορίου μπορεί να συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Και επίσης αναφέρθηκε στον κίνδυνο για τα παιδιά. Είπαν ότι για τα παιδιά είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουν την δόση που ε, ε, με τις δόσεις που υπάρχουν στο νερό στην Ιρλανδία. Και τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφές ε, πλεονέκτημα με την θωρίωση του νερού σε σχέση με την τοπική αγωγή. Και η Επιτροπή ΣΕΡ είπε ότι ε, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι νεότεροι. Διότι αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο να ξεπεράσουν τα, την ε, συνιστόμενη δόση για το φθόριο. Ένα μωρό, εάν ε, λάβει υποκατάστατο μητρικού γάλακτος με... Ε, που ανακατεύεται με νερό θα λάβουν 100 φορές περισσότερο φθόριο από, ότι, ε, από το μητρικό γάλα. Αυτά λοιπόν ε, είπε η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρώπης. Η Ιρλανδία αποτελεί απόδειξη για το πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσει κανείς ε, το όριο. Διότι ε, από τότε που, έγινε, που κρίθηκε παραδεκτή η αναφορά το 2007, περίπου 5.000 15 θα έχουν υποστεί ζημία στο το σμάλτο του, του, των, των, των διών λόγω της έκθεσής τους σε, σε ε, φθοριωμένο ε, νερό. Και ε, τουλάχιστον 10.000 ακόμα θα έχουν επηρεαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί περισσότερο φθόριο από ότι εμείς στην Ιρλανδία. Εμείς μειώσαμε τη δόση. Ωστόσο, τα αποδεκτικά στοιχεία ε, από τη ζημιά που προκαλεί η θωρίωση ε, δεν δημοσιεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και προφανώς για πολιτικούς λόγους. Ε, εφόσον γιατί είναι άγνωστες αυτές οι ζημίες που προκαλεί το φθόριο σε τόσους ανθρώπους. αυτήν ε, την, ε, την γιατί δεν ε, την, τη ζημιά δηλαδή που υφίσταται τα δόντια, γιατί δεν την βλέπουμε στα 436 εκατομμύρια ανθρώπων στο, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ απλό. Η μαζική ιατρική αγωγή με ευθόριο δεν αιτιολογείται. Τα ε, άλλα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι ε, πολύ χοντροκομμένο το μέσο αυτό και δεν ε, αιτιολογείται. Αν τα άλλα κράτη-μέλη εφαρμόζαν το ίδιο, η ευθορίωση στα παιδιά θα αυξανόταν δραματικά και τα και η δοσολογία θα υπερεύαινε την, ε, τα ασφαλή όρια σύμφωνα με την ΕΦΣΑ. Και όσον αφορά τα ιστορικά παραδεκτά αποδεκτά ε, μέτρα, όρια ασφαλείας, ε, το 70% των το 60% των ενηλίκων ε, θα ε, ελάμβαναν ε, περισσότερο φθόριο από ότι η ανώτερη ημερήσια δόση και το 70% των ενηλίκων στην Ιρλανδία. Είναι απόλυτα σαφές λοιπόν το μήνυμα της Επιτροπής σας και θα πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή που δημοσίευσε μία απλή περσιόν των συμπερασμάτων ε, της Επιστημονικής Επιτροπής. Ε, και σας παραθέτω από την έκθεση αυτή. Τι αποτελέσματα είχε αυτό το πολύ σαφές μήνυμα που στέλνουν οι Ευρωπαίοι επιστήμονες. Ε, τι αποτέλεσμα είχε αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανένα απολύτως. Το, το, τον Μάιο του 2011 είδαμε την έκθεση αυτή και μα είπαν ότι αν θέλετε να αλλάξει η πολιτική αυτή, μπορείτε να προσφέρετε στα δικαστήρια. Το οποίο αποτελεί απαράδεκτη απάντηση. Το, το Σάββατο στο Χάμψα έγινε συνάντηση ανθρώπων που εκπροσωπούν κατοίκους, εκ των οποίων 200.000 ε, ε, θα αρχίσουν να λαμβάνουν τώρα φθόριο παρά τη θέλησή τους. Άρχισαν λοιπόν να στέλνουν κάρτες ότι αρνούνται να ε, λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή με το προϊόν αυτό. Ε, αγνοούνται λοιπόν οι κίνδυνοι από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει όμως ε, μια σημαντική πτυχή που είναι η νομική πτυχή αυτής της πρακτικής. Το 1963, όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση είπε ότι όλοι θα πρέπει να λαμβάνουν ε, αυτή αυτή την ουσία στο νερό τους, ε, είπαν ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ε, είδος ε, φθορείου και άρχισαν να χρησιμοποιούν ένα προϊόν το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την παραγωγή λιπασμάτων, το οποίο είναι το φθοριοπυρητικό οξύ. Είχαν λοιπόν μεγάλη παραγωγή λιπασμάτων. Ε, δεν αποτελεί λοιπόν ε, σύμπτωση ότι χρησιμοποιήθηκε ακριβώς αυτό το προϊόν τη συγκεκριμένη στιγμή. Ε, και υπάρχουν πολλά καρκινογόνα, μόλιβος και στην ουσία αυτή και χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα. Όταν ε, συνειδητοποιήσετε λοιπόν από πού προέρχεται το προϊόν αυτό, δεν ε, θα σα εκπλήξει ότι δεν ε, έχει γίνει αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντο αυτού ούτε στην Ιρλανδία ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Παγκόσμιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποσχέθηκε το 2003 ότι ε, θα στείλει μελέτη πάνω στο μόριο αυτό του θωριοπηρητικού οξέως, αλλά ακόμα περιμένουμε την έκθεση αυτή της παγκοσμιου Υγεία. Οργάνωσης Υγείας. άλλα κράτη-μέλη γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα και απορρίπτουν την μαζική φαρμακευτική η αγωγή μέσω του πόσιμου νερού με την χρήση αυτού του προϊόντος. Η δόση είναι αδύνατον να ρυθμιστεί σωστά, ε, συσσωρεύεται στα οστά και ε, προκαλεί μόνιμη βλάβη στα δόντια περίπου ε, του μισού των παιδιών. Ενδιαφέρον είναι να σημειώσει κανείς ότι σε, άλλε, σε άλλα θέματα που αφορούν αξιολογήσεις κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, ε, υπάρχει άμεση ανταπόκριση από την Επιτροπή. Όσον αφορά, για παράδειγμα, ε, τα ε, εμφυτεύματα για τους μαστούς, διότι βρέθηκε εδώ μια μορφή σιλικόνης που φάνηκε ότι πιθανότατα να είναι επικίνδυνη και η Κομισιόν συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ ε, αυξημένη η κίνδυνη σε σχέση με αυτό που πιστεύαν πιο νωρί και γι' αυτό ενέκρινε μια ε, νέα οδηγία 2013-12 που άλλαξε αμέσως το προφίλ κινδύνου της σιλικόνης που χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία PIP. Και ανακάλεσε όλες τις ε, άδειε που είχαν δοθεί για τα υλικά για τα εμφυτεύματα μαστού ε, και είπαν ότι θα πρέπει να επανυποβάλλετε ε, αιτήσει για έγκριση των προϊόντων αυτών προτού να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για φαρμακευτικούς λόγους, για ιατρικού λόγους. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε μεγαλύτερη αντίθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησε αμέσως τον κίνδυνο για τις γυναίκες ε, που ε, είχαν ε, χειρουργηθεί. Όσον αφορά όμως το φθοριοπηρητικό οξύ στο νερό, το οποίο πίνουν όλοι οι Ιρλανδοί και ακόμα και σε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, που το πίνουν ακόμα και, ε, και μωρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα. Ε, σας παρακαλώ να κλείσετε τώρα, λέει η Πρόεδρος, διότι διερμηνία έχουμε ακόμα μόνο για 10 λεπτά. Ε, Ε, ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα, γιατί το βρίσκουν τόσο δύσκολο οι κυβερνήσεις ε, της Ιρλανδία και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ένα προϊόν ε, το οποίο δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει αξιολογηθεί, το οποίο προστίθεται στο νερό, ενώ υπάρχουν ένα σωρό άλλα προϊόντα τα οποία έχουν εγκριθεί και τα οποία χρησιμοποιούνται για τοπική αγωγή και χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και χρησιμοποιούνται ευρέω για την αποφυγή της τεριδόνας. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή σας να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά ε, την νομοθεσία περί φαρμάκων και τροφίμων, η οποία παραβιάζεται με τη φθορίωση του πόσιμου νερού. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία και αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσίασή σα ε, και τώρα εκπρόσωπο τη Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή που ασχολείται με παρόμοια θέματα. Ο κύριος Γιώχεν Ευγένιος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την εισαγωγή. Νομίζω ότι μας έδωσε τη γενική εικόνα. Δεν θα παρουσιάσω λοιπόν και εγώ όλο το ιστορικό, θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον αναφέροντα που μου αντέδρασε θετικά και με την γνωμοδότηση, και στη γνωμοδότηση της, ε, του Συμβουλευτικού Οργάνου γιατί θεωρούμε ότι πράγματι η Επιστημονική Επιτροπή κατέβαλε πολύ καλή προσπάθεια. Θυμούμαστε τότε που κάναμε μια συζήτηση εδώ πέρα για το αν έπρεπε να εξετάσουμε τα επιστημονικά δεδομένα και αν συμφωνούσαμε να ζητήσουμε τη γνωμάτευση της Επιστημονικής Επιτροπής και θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κάνουμε έτσι μια ανοιχτή και διαφανή συζήτηση ε, βεβαίως και χαιρετίζουμε την διαδικασία και με το αποτέλεσμα. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Το σημειώνουμε, κάνουμε μια προσεκτική ανάλυση, όπως και εσείς. Ε, δεν ε, είναι σκόπιμο εδώ να τα κοιτάξουμε γραμμή προς γραμμή όλα τα όσα είπατε. Η κύρια παρατήρησή μου είναι ότι το κύριο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Το τελευταίο σχόλιο του ομιλητή και εμείς και πάλι σε πέρασμα καταλήγουμε. Εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία στον Ηνωμένο Βασίλειο ισχύει, δεν υπάρχει παραβίαση. Βεβαίως, η Επιτροπή, δεν είναι η Επιτροπή που θα πει αν θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική. Εφόσον γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία, εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα ήθελα να σας παραπέμψω και σε μια απάντηση, σε γραπτή ερώτηση του ε, Επιτρόπου Ποτότσνικ το 2011, ερώτημα 4990. Εξετάσαμε και την γνωμάτευση της ε, Επιστημονικής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να δούμε αν έχουμε αρκετά στοιχεία που να δείχνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και όπως απάντησε ο κύριος Ποτότσνικ, η Επιτροπή δεν ε, θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Επικροτούμε αυτή την επιστημονική συζήτηση, θα θέλαμε να συνεχιστεί και να μας ε, παράσχει ε, ενδεχομένω στοιχεία, αλλά σε ό,τι αφορά την νομοθεσία καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν ε, υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας και δεύτερον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αιτιολογούν την αναθεώρηση της νομοθεσίας. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση της θέσης της Επιτροπής. Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Παρακαλώ, Χέλμερ. Παρακαλούμε πώς θα μπορούν να είναι ιδιαίτερα σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Όπως πάντα θα ακολουθήσω ε, τις οδηγίες σας. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πόκοκ για την ε, πολύ καλή του παρουσίαση. Ως σημείο αφετηρία έχω ένα αρνητικό ε, αίσθημα, μια αρνητική εντύπωση όταν λέμε ότι θα πρέπει να ε, χορηγήσουμε κάποιο είδους αγωγή στον πληθυσμό χωρίς ε, την ε, σύμφωνη γνώμη τους. Γι' αυτό και δεν θέλω να υπάρχει φαρμακευτική αγωγή στο, στο πόσιμο νερό, εκτός και αν υπάρχει κάποια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Αλλά αυτό δεν ισχύει εδώ. ο ο αναφέρον ε, μίλησε για ζημιά στα δόντια λόγω της υπερβολικής θεωρίας του νερού. Εγώ σήμερα έλαβα ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ιρλανδία. Είναι κάτι που συνεχίζεται, δεν το είχα εξετάσει ε, Και εκεί φαινόταν ότι τα τρέχοντα επίπεδα φθορίωσης προκαλούν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και προβλημάτων πέρα από τα δόντια. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δεν είμαι ειδικό ε, επί του θέματο, αλλά μου φαίνεται λογικό. Υπάρχουν επιχειρήματα, και ιδιαίτερα αρνητικά επιχειρήματα, Ω ε, ευρωσκεπτικιστή χαίρομαι που η Επιτροπή δεν προτείνει να ε, παρέμβει στα αρμοδιότητε των κρατών μελών. Όμω για το αν θα πρέπει να υπάρχει φθοριώση του νερού, εγώ έχω αρνητική στάση. Και μετά τα όσα άκουσα και σήμερα το πρωί, είμαι ακόμα πιο αρνητικό από ό,τι ήμουν στην αρχή. Σα ευχαριστούμε και εσά. Μάρφη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την ε, παρουσίασή του. Ήταν ιδιαίτερα σαφής. Είναι προφανώ ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα κατά τη φθορίωση ό,τι αφορά του κινδύνου για την υγεία. Βεβαίω και για την οδοντική φθορίωση και για τα υπόλοιπα όμω. Περιβαλλοντικέ επιπτώσει, η διαρροή ε, ποθέματα ε, αποθέματα νερού αλλά και αλλού. Όπως αναφέρει και η Επιτροπή, πράγματι δεν είναι σημαντικά τα ωφέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η αρχή της πρόληψης, αυτή να ισχύει εδώ, και να μην ε, εισάγουμε ευθόριο στο νερό. Αλλά υπάρχει και ένα δημοκρατικό ζήτημα. Το δικαίωμα το, μιας κοινότητας να μην ε, λαμβάνει μια ουσία αν δεν το επιθυμεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί δεν υπήρξε ευρύς διάλογος ε, και με δημοκρατικές ε, διαδικασίες να αποφάσισε ο πληθυσμό ε, να εισαχθεί το φθόριο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό η Επιτροπή ε, η συγκεκριμένη Επιτροπή να εξακολουθήσει να ασκεί πιέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ιρλανδική κυβέρνηση να αποσύρει το φθόριο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Ρόμπερτ Βόκακ. Ήμουν εδώ την τελευταία φορά που το παρουσίασε και τον στηρίζω εξ αρχής. Τρεις ε, παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, η Επιτροπή στην απάντησή της είπε ότι δεν πιστεύει ότι το φθόριο μπορεί να θεωρηθεί ε, φαρμακευτική ουσία. Αλλά το ερώτημα μου είναι γιατί το προσθέτουν τα κράτη-μέλη στο νερό. Γιατί αν κάτι είναι φαρμακευτική ουσία, είτε ε, θεραπεύει, είτε αποτρέπει παθήσεις. Τα κράτη-μέλη το προσθέτουν γιατί αποτρέπουν έτσι την τεριδόνα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Η Επιτροπή είπε πριν, πριν από λίγο ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να, που αιτιολογούν μεταρρύθμιση, αναθεώρηση της νομοθεσίας. Εγώ ε, κοίταξα την Επιτροπή Σέρφτη και τα συμπεράσματά της για μένα είναι επαρκή ε, για την επανεξέταση της νομοθεσία από την Επιτροπή. Γιατί σύμφωνα με την έκθεση υπάρχει κίνδυνος ε, οδοντικής για τα παιδιά και ότι δεν υπάρχει ανακατόφλη. Μιλάει για, έν για ανώτατο επίπεδο. Όχι για χαμηλότερο, ανώτερο επίπεδο. Και λέει συγκεκριμένα και παραθέτω ότι επιτύχεται, επιτυχάνεται σε παιδιά 6 έως 10 ετών που μένουν σε αυτή την περιοχή και πίνουν πάνω από ένα λίτρο νερό και χρησιμοποιούν ε, την ε, οδοντόπαστα που περιέχει φθόριο και η ποσότητα και πέρα είναι όσο ένα μπιζέλι, έτσι, να το έχουμε αυτό κατά νου. Και σε αυτή την περίπτωση των παιδιών 6 έως 12 ετών ξεπερνούν ε, κατά πολύ αυτό το, αυτό το όριο. Και για τα παιδιά από 1 έως 6 ετών, αν πίνουν μισό λίτρο νερό και χρησιμοποιούν αυτήν την οδοντόπαστα με το φθόριο, και πάλι υπερβαίνεται το ανώτερο επίπεδο. Ε, και για τα βρέφη κάτω των 12 μηνών, Διαφωνώ εδώ με τους αναφέροντες. Είπε ότι η έκθεση στο φθόριο είναι 100 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το μητρικό γάλα. Όχι, είναι 200 φορές ε, μεγαλύτερη έκθεση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, λέω λοιπόν στην Επιτροπή ότι εφόσον έχουμε αυτά τα αποτελέσματα από την έκθεση share, σίγουρα υπάρχουν ε, στοιχεία. Τώρα, αν είναι επαρκή ή όχι, εγώ πιστεύω πω είναι. Αλλά υπάρχουν στοιχεία που αιτιολογούν την επανεξέταση του ζητήματο. Και τέλο, έχουμε σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, βιοιατρική. Πολλοί το έχουν υπογράψει, Δανία, Ελλάδα, Κύπρος, ε, Βουλγαρία, σχεδόν 20 χώρε το έχουν υπογράψει και κυρώσει. Δύο χώρε μόνο δεν το έχουν κάνει, ε, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Και σίγουρα ένα από του λόγου είναι το γεγονό ότι προσθέτουν φθόριο στο νερό. Το άρθρο 5 της σύμβασης λέει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση υγειονομική μπορεί να γίνει μόνο μετά από ε, τη σύμφωνη γνώμη ε, και διαβούλευση με και σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Εγώ λοιπόν προτείνω στην Επιτροπή Λέω στην Επιτροπή ότι ε, η, η έκθεση ΣΕΡ παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ε, επανεξέταση της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να παρακαλέσουμε την Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να ε, δώσει τέλος σε αυτήν την ε, κατάσταση. Ε, εμένα αυτά μου θυμίζουν σοσιαλισμό, μου θυμίζουν τα νιάτα μου στην Ανατολική Γερμανία όπου δεν μπορούσε να ρωτήσει κανείς το κράτος τι, τι, προσμίξεις γινόντουσαν. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται, διότι το πόσιμο νερό είναι διαθέσιμο σε όλου. Ε, δεν μπορεί λοιπόν κανεί να βάλει ό,τι θέλει στο πόσιμο νερό. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο στην ιστορία αυτή. Εγώ όταν αγοράζω κάτι στο σούπερ μάρκετ ή στο φαρμακείο, ξέρω τι αγοράζω. Μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Έχουμε την οδηγία για το πόσιμο νερό, έχουμε διάφορες προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμένα με ενοχλούν αυτές οι προσμίξεις, είτε θεωρείτε ότι είναι φαρμακές ή όχι. Όσον αφορά άλλα ανώτατα όρια, είμαστε πιο προσεκτικοί. Πιστεύω λοιπόν ε, ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους αναφέροντες. Κάτι εδώ δεν πάει καλά και θα πρέπει η Κομισιόν ε, να το εξετάσει. Εμεί ω Επιτροπή Αναφορών ε, θα ε, συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και θα αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή εάν έχει πολύ σύντομα κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρεμβάσεις. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι δεν είναι ερμηνεία της Κομισιόν ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Βασιζόμαστε σε συμπεράσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και, τα, και τις αναθεωρημένες κατευθυντήρες που δημοσιεύτηκαν πέρσι και έχουν συζητήσει όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στην έκθεση της ΣΕΡ. Είμαστε συνεπείς λοιπόν με τις κατευθυντήρες γραμμές και τις... Ε, εάν υπάρχουν νέα επιστημονικά στοιχεία, διότι τα επιστημονικά στοιχεία εξελίσσονται συνέχεια και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία καταλήξει ότι έχει αλλάξει η κατάσταση, τότε εντάξει. Αλλά γι' αυτό έχουμε φτάσει ε, σε ένα ε, σημείο που δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την ε, οδηγία για το πόσιμο νερό. Αυτό το μόνο είχα να προσθέσω. Σα ευχαριστώ όλου πάρα πολύ. Και για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης ε, της συναντησής μας. Ε, να σας πω ότι λάβαμε υπόψη μας, σημειώσαμε... Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, αναφέρον θέλει κάτι να πει. Συγγνώμη, δεν έχω το δικαίωμα να απαντήσω στην απάντηση της Επιτροπής. Ε, this reunion, is... Έχουμε φτάσει στο τέλος της συνεδρίασης κανονικά τελειώνουμε στις 12.30 και οι, οι θα φύγουν. Ναι, αλλά αξιοποιήσατε το χρόνο σας ε, σήμερα το πρωί. Εντάξει, πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να απαντήσω. Θα ήθελα... Η Πρόεδρος λέει ότι εξ αρχής ε, μακρηγορήσατε, γι' αυτό δεν σας έδωσα επιπλέον ε, λόγο αν έχετε κάτι πολύ σύντομα να προσθέσετε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, εκπροσώπους από τα άλλα κάτι μέλη που αναγνωρίζουν το σημαντικό πρόβλημα ε,